Good morning, Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε νωρίς σήμερα το πρωί γιατί έχουμε πάρα πολλά στην ημερήσια διάταξη. Σας παρακαλώ καθίστε και σας ευχαριστώ που ήρθατε και στην ώρα σας όσοι ήρθατε στην ώρα σας. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης, σημείο 1. Έχουμε τις εξής αλλαγές. Ε, το σημείο 7 σε ό,τι αφορά την ε, αποστολή στην Τουρκία αναβλήθη σε ό,τι αφορά το σημείο 14 στις 2 αντί για τις 2.45, το 15 για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, η παρουσίαση της ενδιάμεσης αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Προσθέμενης Αξίας στις 3, ε, πριν από το 14. Αν δεν έχετε αντιρρήσει, εγκρίνονται. Um, I I to... Και τώρα περνάμε στι ανακοινώσει του Πρόεδρου. Καταρχά, ό,τι αφορά τι γλώσσε. Και πάλι δυστυχώ δεν έχουμε τα κρατικά και τα ελλανδέζικα. Να σα υπενθυμίσω ότι στι 10.45 έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. σα παρακαλώ να έχετε τι κάρτε σα. Συνάδελφοι, για όσους έχετε έρθει στην ώρα σας. Θα ξεκινήσω και δεν θα σας προκαλέσει έκπληξη ότι θα ξεκινήσω την πρώτη συνεδρία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, η οποία είναι και η πρώτη μετά τις τρομερές τρομοκρατικές επιθέσεις στις 22 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, με δύο λόγια για τα περιστατικά αυτά. Ήταν και έκτακτη, είχαμε και την έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υπουργών Ιστορικών στις, ε, μετά τις επιθέσεις και θα ήθελα να πω δύο λόγια και για αυτή τη σύνοδο. Να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Ιγουγιών να μας ε, ε, δώσει, να μας παρουσιάσει το τι έγινε και τι εκπροσώπησε το Κοινοβούλιο στη συνάντηση αυτή. Όπως σας είπα, είναι η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έχει και φέρει μια ιδιαίτερη ευθύνη σε ό,τι αφορά το τομέα αυτό. Πάνω από 30 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 240 άτομα τραυματίστηκαν. Και φυσικά θέλουμε να αποτίσουμε φόρο του εμείς στα θύματα, στις οικογένειές τους, στους Βέλγους πολιτές και ασφαλώς ε, και στα, στους ηθήνοντες και στις αρχές του Βελγίου. Τρεις μέρες εθνικού πένθους ανακηρύχθηκαν στο Βέλγιο και αυτό ισχύει και για όλους τους Ευρωπαίους ουσιαστικά. Θα συμφωνείτε, φαντάζομαι, μαζί, μαζί μου ότι εκφράζουμε την ε, συμπόνια μας και την αλληλεγγύη μας προς όλους τους Βέλγους. Και εξ ονόματος της Επιτροπής μας θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Thank you, colleagues. So, colleagues, um... Συναδελφοί, λοιπόν, στην πρώτη συνέδρια λοιπόν, τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ μετά τι τρομοκρατικέ επιθέσει, είναι σημαντικό, ε, θεωρώ, να πούμε προς το κοινό που παρακολουθεί την συνεδρίαση της Επιτροπής και στα μέλη μας, τα οποία αντιδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε όλα τα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι Χρειαζόμαστε μια μεγάλη σειρά μέτρων για να καταπολεμήσουμε τις διάφορες διστάσεις τη τρομοκρατίας ε, σε δικαστική και αστυνομική συνεργασία, ε, κοινή αξιοποίηση των πληροφοριών, καταπολέμηση της παστικοποίηση σε ό,τι αφορά την εκτεστάτε και πάρα πολλά πολλές άλλες πτυχές της εργασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και πρέπει να σας πούμε ότι δεν βρισκόμαστε ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο σε ό,τι αφορά την κοινή αξιοποίηση των πληροφοριών και τα κράτη-μέλη ασφαλώς πρώτα θα, πρέπει να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα σε ό,τι αφορά το SIS, το σύστημα SIS και άλλες ε, διακυβερνητικέ αποφάσει για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και την ανταλλαγή δεδομένων. Καλό λοιπόν την Επιτροπή, εξ ονόματο τη δική μα Επιτροπή, να εξασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη τα οποία ακόμα δεν έχουν χορηγήσει τα απαραίτητα δεδομένα θα εφαρμόσουν τις αποφάσεις αυτές ε, τις οποίες ακόμα δεν έχουν εφαρμόσει. Και μάλιστα μερικές εξ αυτών ε, είναι και το 2008 έχουν περάσει. Και νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό, συναδελφοί, ακριβώς για τους πολίτες που παρακολουθούν τη συνεδρίαση, να κατανοήσουμε ότι η Επιτροπή μας και τα μέλη μας ε, εργάζονται για το σύστημα ΕΚΡΙΣ σε ό,τι αφορά την έκθεση Κέρκοπ για τους ε, υπηκόους ε, τρίτων χωρών και σε ό,τι αφορά επίσης τα εξωτερικά σύνορα και έκθεση Μάκοβη, ε, οδηγία Χόλμα για την έκθεση Χόλμαϊερ και όλα αυτά τα οποία αποτελούν τα απαραίτητα νομοθετικά εργαλεία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτές είναι μερικές ορισμένες, ορισμένες μόνο πτυχές της Αντρέντα για την ασφάλεια που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητάς μας σε ό,τι αφορά και τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Είπα λοιπόν συνάδελφοι στην αρχή τη ανακοινώση ότι στι 24 Μαρτίου μετά τι τρομοκρατικέ επιθέσει, οι Υπουργοί Δικαιοσύνη συναντήθηκαν για να συνομιλήσουν και να, συναντήσουν την, να συζητήσουν την κατάσταση για τις επιθέσεις και είχαμε την κυρία Κουγιώνα εκπρόσωπο της Επιτροπής μας στην συνάντηση αυτή και θα ήθελα να μας δώσει τώρα μια σύντομη παρουσίαση της συνάντησης εκείνης. Ε, δεν ε, έχουμε πολύ χρόνο, θα πάρει το λόγο και θα μας μιλήσει ε, εν συντομία Σιλβία, αν θέλεις, πάρει το λόγο. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε όντως ότι αντιπροσώπευα το Κοινοβούλιο και ε, όντως ε, συμφωνώ με τα όσα είπατε απολύτως. Η παρουσία μου σε αυτήν ε, την σύσκεψη του Συμβουλίου ήταν να διευκρινίσω και να εκφράσω τη στήριξη του θεσμού που αντιπροσώπευα εκείνη την ημέρα σε σχέση με τις επιθέσεις που χτύπησαν το Βέλγιο πριν λίγες μέρες από εκεί την εξαγωγή εκείνου του Συμβουλίου και επίσης να πω τι θέλουμε να ενισχύσουμε στη βάση της δημοσίευσης της ατζέντα σε σχέση με την ασφάλεια με, από πλευρά των Κομισιόν ε, μπορέσαμε να μιλήσουμε και να αξιολογήσουμε το την ανάγκη να προχωρήσουμε, να καταπολεμήσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση και άλλα σημεία τα οποία δεν θέλω να επαναλάβω. Απλά να πω δύο λόγια σε σχέση με συμπληρωματικά με τα όσα είπατε. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να υπογραμμίσουμε τα κρίσιμα σημεία ε, της ανταλλαγής των πληροφοριών που ξέρετε πολύ σχολιάζεται με παρεμβάσεις ε, σε σχέση με την διαλειτουργικότητα, την ανάλυση δεδομένων που έχουμε, καθώς και τους πόρους που μοιραζόμαστε. Είναι ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε και ευχαριστώ και σύντομα ακριβώς σας έκανα την έκθεσή μου για αυτό το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ Σιλβή και όπως είπες είναι ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθουμε. Ξέρω πως πολλοί θέλουν να το συζητήσουμε, αλλά δεν έχουμε το χρόνο να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό θα, ε, ήθελα να συζητήσουμε ε, να συζητήσουμε το ενδεχόμενο να καλέσουμε τον κύριο Γιάννη Γιάνν Μπον, τον Υπουργό Εσωτερικών του Βελγίου, να έρθει εδώ, αλλά και τον Υπουργό της, ε, που είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου, κύριος Κουν Χένς, ε, εδώ, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Επίσης θα πρέπει να ακούσουμε τον, Ευρωπαϊκό, τον Ευρωπαίο Συντονιστή της Europol για, για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Στην επόμενη λοιπόν ε, εβδομάδα θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τους συντονιστές. Ε, προχωράμε λοιπόν στο σημείο 3 με 6 που είναι οι διάφορες παρουσιάσεις από την Κομισιόν και τα διάφορα ανακοινοθέντα που μας έχουν απασχολήσει σε σχέση με την Ένωση Τουρκία και, και, την ε, συνεργασία με την Τουρκία για το μεταναστευτικό. Θα προχωρήσουμε γρήγορα γιατί έχουμε λίγο χρόνο για κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλους μας στην Επιτροπή. Η μεταναστευτική κρίση βεβαίως έχει οδηγήσει σε πολύ στενότερη και εντατική συνεργασία με την Τουρκία για θέματα μετανάστευσης. Είδαμε όλες τις εξελίξεις τελευταίες μέρες. Έχουμε διάφορες λοιπόν πτυχές που θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα και θέματα κυρίως ε, επιχειρησιακά, αλλά δεν θα περιοριστούμε σε αυτά μόνο. Η Επιτροπή βεβαίω έστειλε, την έστειλε αντιπροσωπεία στην Τουρκία και συμβάλαμε με μια τακτική έκθεση, για σε μια τακτική έκθεση μάλλον της για την Τουρκία στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Τώρα θα ήθελα βεβαίω να συζητήσουμε και να εστιάσουμε περισσότερο στο τι αναμένουμε από την Κομισιόν Βεβαίω και από τα κράτη-μέλη και γι' αυτό το λόγο Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Μάρτιν Βερβέ, που όσοι δεν το γνωρίζετε ακόμα, ορίστηκε από τον πρόεδρο Γιούνκερ να, ώστε να λειτουργήσει ως συντονιστή για να εφαρμοστεί η Συμφωνία Ένωσης με Τουρκία. Εκείνο λοιπόν πρέπει να ακούσουμε. Είναι υπεύθυνο για τα επιχειρησιακά ζητήματα. Θα προβεί σε μια σύντομη δήλωση. Έχουμε και άλλους συναδέλφους εδώ από την Επιτροπή. Ε, και θα ήθελα να εστιάσουμε την προσοχή μας λοιπόν σε αυτή την εισήγηση και μετά να δούμε ερωτήσεις ε, ή απορίες για αυτό το πολύ σημαντικό ε, θέμα. πολύ ε, χαιρόμαστε λοιπόν που είστε κύριε Βερβέη εδώ σήμερα και σας δίνω το λόγο για να ξεκινήσετε την εισήγησή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή σας που με δέχτηκε σήμερα. Θα ήθελα να σας κάνω μια ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις από τις 18 ε, Μαρτίου μέχρι σήμερα, όταν δηλαδή ανακοινώθηκε η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Το έργο μου είναι ο συντονισμός όλων των ε, επιχειρησιακών προσπαθειών για την εφαρμογή αυτής της δήλωσης. Πριν όμως θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τι ε, έγραφε η δήλωση. Πιστεύω πως ε, κεντρικό θέμα της συμφωνίας είναι το εξής, τα εξής δύο μάλλον. Η Τουρκία δηλαδή δεσμεύτηκε να πάρει πίσω όλους τους παράτυπους μετανάστες οι οποίοι πέρασαν από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά από τις 20 Μαρτίου. Και έπειτα για κάθε Σύριο που επιστρέφει στην Ελλάδα, δύο, ε, που επιστρέφεται από την Ελλάδα, δύο θα απορροφούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε λοιπόν μια δέσμευση επίσης για την επίσπευση του, της ε, απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρέχει χρηματοδότηση για να βελτιωθούν οι συνθήκες ε, στην Τουρκία για τους μετανάστες. Όπως ε, επίσης γνωρίζετε υπάρχουν αναφορές στα αντίστοιχα κεφάλαια διαπραγματεύσεων ε, για την ένταξη της Τουρκίας. Στόχος όλων αυτών είναι να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το επικίνδυνο πέρασμα από το Αιγαίο να σταματήσει ε, αυτή η διακίνηση από τους ε, διακινητές στην Τουρκία και να γίνει σεβαστό το διεθνές ε, και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Τι έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Ας δούμε καταρχάς κάποιους αριθμούς. Εδώ βλέπουμε πραγματικά αποτελέσματα. τον μήνα πριν την συμφωνία οι ημερήσιες αφήξεις στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 1676 την ημέρα. Τώρα ο ρυθμός αυτός έχει μειωθεί στους 399 κάθε μέρα. Αυτήν την εβδομάδα είδαμε μία ακόμα μείωση. Προχθές 68 άνθρωποι έφτασαν στην Ελλάδα και την προηγούμενη ε, μέρα 76. Ένα από τα αποτελέσματα, μάλλον ένας από τους ε, στόχους όλου αυτού είναι το εξής. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 21η Μαρτίου Δηλαδή, μέχρι να παρατηρηθεί αυτή η μείωση στις αφήξεις, 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Από τις 21 Μαρτίου μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει χάσει τη ζωή του. Αυτό φυσικά δεν καθιστά πρόβλεψη για το μέλλον, όμως είναι μια λογική ε, συνέπεια της μείωσης του αριθμού των ε, ανθρώπων που καταφθάνουν. Σίγουρα πολλά πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να είναι υλοποιήσιμη η συμφωνία αυτή και να διασφαλιστεί ότι όντως το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο γίνεται σεβαστό. Και έχουν ήδη γίνει αρκετά. Καταρχάς υπάρχει συμφωνία, επιχειρησιακή συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας για την έπαν ιστοχή. Υπάρχουν σύνδεσμοι στην, ε, της Ελλάδας στην Τουρκία και το αντίστροφο. Έχουν γίνει αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο. για την εφαρμογή της πρώτης ασφαλούς χώρας ε, εισόδου για όσους ετούνται άσυλο και για την ε, δήλωση της ε, Τουρκίας ε, ως ασφαλής χώρα. Έχει δηλαδή να αλλάξει η νομοθεσία έτσι ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις πεσμένες διαδικασίες. Θεωρείται δηλαδή η χώρα ασφαλής. Και υπάρχει δυνατότητα να μην γίνονται αποδεκτά ε, αιτήματα ασύλου. Σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Τουρκίας υπέγραψε μία αλλαγή στην ε, τουρκική νομοθεσία που αφορά τους Σύρους. Αυτό, όπω σα είπα, θα έχει κάποια αποτελέσματα. Δεν έχω δει ακόμα το κείμενο, όμως αναμένουμε να έχει αποτέλεσμα για τους σύρου οι οποίοι επιστρέφουν στην Τουρκία. Εκείνοι θα λάβουν καθεστώ προσωρινή προστασίας, το οποίο μεταξύ άλλων θα τους δίνει πρόσβαση στις ε, αναγκαίες ε, υπηρεσίες αλλά και στην αγορά εργασίας κτλ. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο των συζητήσεων. Φυσικά δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη. Συζητούνται ακόμα αρκετά θέματα σε άλλους ε, τομείς, όμως είναι η πρόοδος που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Επίσης, κινητοποίηση πόρων. Είναι μια μεγάλη επιχείρηση. Η Frontex έχει ζητήσει αύξηση του προσωπικού και μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη έχουν υποσχεθεί 730, 736 υπαλλήλου για να προσθεθούν στους 263 που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ελληνικά νησιά. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου επίσης έχει λάβει την υπόσχεση από τα κράτη-μέλη για 452 πρόσθετους υπαλλήλους. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει πρώτη ομάδα υπαλλήλων της ΕΑΣΟ, 30 υπάλληλοι και διερμηνείς, οι οποίοι έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται αυτά τα αιτήματα ασύλου. Επίσης, όπως γνωρίζετε, έχουν ήδη αρχίσει ε, οι πρώτες ε, εξέργασης συστημάτων ασύλου. 74 Σύρι μέχρι τώρα θα κατασταθούν από την Τουρκία σε τρία κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω πως σε γενικές γραμμές έχουν κυλήσει ομαλιά αυτά μέχρι τώρα. Σίγουρα υπάρχουν προκλήσεις και μάλιστα αρκετές. όπως άλλωστε είναι φυσικό σε μια επιχείρηση τέτοιου μεγέθους. Όμως έργο μας είναι, μέσω των προκλήσεων αυτών, να καταφέρουμε όλα τα αιτήματα ασύλου που έχουν εισαχθεί στο σύστημα να επεξεργαστούν κατά περίπτωση σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό φυσικά προϋποθέτει την αύξηση των ε, ικανοτήτων ασύλου Και επίσης να πω ότι μας απασχολούν οι συνθήκες ε, στα κέντρα υποδοχής, στα hot spots. Ακόμα και τις πρώτες μέρες που ε, παρατηρήθηκε αυτή η μείωση υπήρχε προσέλευση. Και αυτή τη στιγμή τα hot spot είναι υπερφορτωμένα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τις αρχές έτσι ώστε να αυξήσουμε πάρα πολύ γρήγορα τη χωρητικότητα. Επίσης υπήρχε ένα πρόβλημα στην παροχή υπηρεσιών, υπήρχε έλλειψη παροχής υπηρεσιών και αυτό γιατί ήταν πάρα πολλές ΜΚΟ που παρήχαν αυτές τις υπηρεσίες και σταμάτησαν να το κάνουν για διάφορους λόγους. Εμείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δώσαμε ε, βοήθεια στις ελληνικές αρχές και αυτή η βοήθεια ήταν η ιατρική, ήταν υπηρεσίες catering και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στον τομέα αυτό έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι μετά από αυτό το στάδιο επανακατάστασης πρέπει να δημιουργηθεί μια μόνιμη διαδικασία από την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστροφο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν ασφαλείς οδοί εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, για όσους έφτασαν πριν για όσους φτάσουν πριν τις 20 ε, Απριλίου, που είναι αρκετοί, πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαμονής και να επισπεύσουμε το πρόγραμμα επανεγκατάστασης έτσι ώστε να οδηγηθούν σε ασφαλή ε, μέρος, ασφαλές μέρος. Σας ευχαριστώ και ασφαλώς πολλοί συνάδελφοι θέλουν να, θέσουν ερωτήσεις. Μιλήσατε για αριθμητικά στοιχεία όμως. Να ελέγξω ότι μιλήσατε ε, για κάποιες υποσχέσεις για προσωπικό στην ΕΑΣΟ. Αυτό ισχύει ακόμα. 30, κοιτάξτε, ναι, 32 εμπειρογνώμονες. Συν 30 διερμηνείς. Πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, πρέπει πολύ απλά να υπάρχει και μια εκπαίδευση, μια κατάρτιση. Δεν μπορούμε απλά να αποστέλνουμε ομάδες ε, ατόμων. Θα πρέπει να υπάρχει μια κατάρτιση προκειμένου να υπάρχει ίδιος τρόπος αντιμετώπισης των αιτήσεων ε, για άτομα που είναι από άλλες χώρες και έχουν άλλες πρακτικές, ακολουθούν άλλες πρακτικές. Άρα, σε πρώτη φάση έχουμε ένα πλωτικό πρόγραμμα με περιορισμένο αριθμό ατόμων και στην επόμενη φάση θα υπάρξει αύξηση σταδιακή των ε, ατόμων αυτών. Και θα ακολουθήσουν και άλλες φάσεις ασφαλώς. Συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό και έχω προβλέψει χρόνο για να το συζητήσουμε. Ίσως να έχουμε και χρόνο και για παραπάνω από ένα γύρο. Να ξεκινήσουμε με τους συντονιστές. Η κυρία Βόζεμπεργκ από το ΕΛΚ. Θα πάρετε το λόγο κυρία Βόζεμπεργκ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βερβέη που ήρθε να μας ενημερώσει για τα πρώτα στάδια της εφαρμογής της συμφωνίας ε, κύριε Βεβέη, προέρχομαι από την Ελλάδα και καταλαβαίνετε ότι είναι η πρώτη χώρα που βιώνει με δραματικές ε, εκτάσεις το πρόβλημα αυτό. Θέλω να σας ενημερώσω ότι καταρχάς γνωρίζετε ότι για την Ελλάδα η Τουρκία δεν έχει αναγνωριστεί ως ασφαλής χώρα. Με συνέπεια, σύμφωνα με τον νόμο, όσοι ζητούν άσυλο να παραμένουν μέχρι να κριθεί το αίτημά τους στη χώρα μας. Τι έγινε λοιπόν, αμέσως μετά την εφαρμογή της συμφωνίας, την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, όλοι, μπορώ να σας πω, 95% όλων των ανθρώπων που βρίσκονται, των απελπισμένων αυτών ανθρώπων στη χώρα μου, είτε έχουν την ιδιότητα του πρόσφυγα, είτε του παράτυπου μετανάστη, όλοι ζήτησαν άσυλο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εντός 15 ημερών, 14 κατά πρέπει να έχει κριθεί η αίτησή τους, αλλά έχουν δικαίωμα να προσφύγουν σε δεύτερο βαθμό κρίσης, στην Επιτροπή δεύτερου βαθμού κρίσης πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αναγκαστικά οι άνθρωποι αυτοί θα μείνουν στην Ελλάδα. Ούτε έχουμε δικαίωμα να τους στείλουμε πίσω στην Τουρκία, ούτε ώστε εκείνη να τηρήσει τη συμφωνία επανεισδοχής, ούτε μπορούμε ε, να τους διαχειριστούμε διαφορετικά. Το λέω αυτό διότι επιπρόσθετα ξέρετε πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν έχει ένα δεσμευτικό μηχανισμό για τη μετεγκατάσταση. Με άλλα λόγια, και εκεί που θέλουν οι άνθρωποι αυτοί να μεταβούν, έχουν κλείσει οι διάδρομοι, κράτη-μέλη δεν δέχονται να υλοποιήσουν τις αποφάσεις για μετεγκατάσταση και αυτό σημαίνει ότι αναγκαστικά οι άνθρωποι αυτοί θα παραμείνουν στην Ελλάδα. Σε ό,τι μας, ε, αναφέρατε σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας για τα ρεύματα των ανθρώπων που έρχονται από την Τουρκία, να σας ε, ενημερώσουμε και το γνωρίζετε ότι από τις 20 του μηνός που το, άρχισε να εφαρμόζεται τη συμφωνία, οι ροές δεν σταμάτησαν καθόλου. Είναι πράγματι μειωμένες τώρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πλήρη εφαρμογή από πλευράς της Τουρκίας ως συμβαλόμενου μέρους στη συμφωνία. Επιπρόσθετα, δεν έχουμε δει να γίνονται ε, ουσιαστικές κινήσεις από τον έλεγχο των διακινητών για τους οποίους έχει απόλυτη γνώση η Τουρκία και μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει τίποτα. Η ερώτησή μου προς εσάς παρακαλώ είναι ότι εφόσον κατά την άποψη τη δική μου ή τη δική μας η συμφωνία δεν εφαρμόζεται όπως θα έπρεπε να εφαρμόζεται. Μέχρι στιγμής δεν είναι τα αποτελέσματα ικανοποιητικά. Δεν θέλω να πω ότι έχει αποτύχει, απέφχομαι να αποτύχει, αλλά σίγουρα δεν είναι ικανοποιητικά. Προβλέπετε κάποια εναλλακτική ε, λύση για την ε, διευθέτηση του θέματος. Επαναλαμβάνω ότι λόγω του ότι ζητούν όλοι άσυλο και είμαστε υποχρεωμένοι και να το εξετάσουμε στις προθεσμίες που υπάρχουν από τον νόμο. Αλλά και εκείνοι έχουν δικαίωμα να προσφύγουν, ούτω ώστε εκ των πραγμάτων θα παραμείνουν μεγάλο χρονικό διάστημα και επίσης οι ροές δεν έχουν σταματήσει τελείως, απλώς έχουν μειωθεί. Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλο πρόβλημα διαχείρισης από τη χώρα μου, αν λάβετε υπόψη σας επιπρόσθετα ότι είναι η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται σε καθεστώς ε, ε, τήρησης του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Um, for the Σας ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Η κυρία Σίπελ έχει το λόγο. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από την ε, δήλωση αυτή που αποφασίστηκε. Νομίζω ότι πολλοί, παρά την κριτική που είχε ασκηθεί για την Κριτία, την Τουρκία, είχαν την ελπίδα ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε, να, να πετύχουμε μια συμφωνία η οποία στο θέμα των προσφύγων θα έβαζε μία τάξη στο σύστημα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των προσφύγων στην ε, Ευρώπη. και με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να πιστούν και τα κράτη-μέλη που ως τώρα, να το πω προσεκτικά, ήταν κάπως ε, διστακτικά να υποδεχτούν πρόσφυγες. Και κοιτώντα τελικά αυτά που ε, συμφωνήθηκαν και αυτά που διαφαίνονται προς το παρόν, έχω μεγάλες αμφιβολίες. Η εντύπωση που μας δίδεται είναι η εξή ότι γίνεται, μάλλον το μήνυμα που αποστέλλεται είναι ότι πρόσφυγες μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, αλλά να μην έρθετε στην Ευρώπη, γιατί πολλά κρατημέλη δεν είναι διατεθειμένα να υποδεχτούν πρόσφυγες. Και τι άλλο προστίθεται, ότι αν πιστεύουμε ότι όλοι οι πρόσφυγες σε χώρες, θα πρέπει να μείνουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει τουλάχιστον, μα τουλάχιστον, αφού έχουμε δώσει τόσα χρήματα για να σώσουμε τις τράπεζες, να βάλουμε το χέρι στην τσέπη και να υποστηρίξουμε τις χώρες που είναι σαφώς πιο ασταθή και οικονομικά πιο ασταθή από ότι οι δικές μας χώρες προκειμένου να μπορούν να υποδεχτούν πρόσφυγες. Δεν μπορώ πια να ακούω να λένε ότι θέλουμε να μειώσουμε του αριθμού των προσφύγων, μα δεν κάνουμε αυτό. Αυτό που κάνουμε είναι να μειώνουμε τον αριθμό των προσφύγων που έρχονται σε εμά. Α είμαστε ειλικρινεί και ανοιχτοί. Μία ερώτηση όμω έχω να κάνω προ την Κομισιόν, ή μάλλον και πιο πολλέ ερωτήσει έχω να κάνω. Καταρχά, καταρχάς, είπατε ότι η Τουρκία για κάποιε ομάδε ανθρώπων είναι ασφαλή. Μα ποιες είναι αυτές οι ομάδες. Για πείτε μας ποιε θα μπορούσαν να είναι αυτέ οι ομάδες. Δεύτερη ερώτηση. Με νομοθετικέ αλλαγέ στην Τουρκία οι Σύριοι υποτίθεται ότι θα μπορούν να έχουν και να απολαμβάνουν την ε, προστασία που χρειάζονται. Τι γίνεται όμως με τους πρόσφυγες από άλλες χώρες, οι οποίες, με πρόσφυγες από άλλες χώρες, οι οποίοι θα ερχόντουσαν στην Ευρώπη και θα βρεθούν στην Τουρκία. Αυτοί δεν θα προστατεύονται σωστά. Μιλήσατε για επανεκατάσταση. Τρία κράτη έχουν υποδεχτεί ε, πρόσφυγες. Φαντάζομαι ότι δεν πρόκειται για το Ηνωμένο την Δανία, την ε, Πολωνία, τη Γαλλία. Πείτε μας, σας παρακαλώ, ποιες χώρες είναι αυτές. Τρίτον, μας μιλήσατε για 72.000 άτομα από την Τουρκία, τα οποία θα πρέπει να τα υποδεχτούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω καν να συζητήσω τον αριθμό αυτό. Αλλά για τι χρονική περίοδο μιλάμε, για ένα μήνα, για ένα χρόνο, για πάντα. Με τι χρονικό ορίζοντα μιλάμε. Γιατί είναι σημαντικό το ερώτημα αυτό. Και ύστερα θα ήθελα να ξέρω το εξή, να μου πείτε το εξή, για το θέμα της ε, σχολικής εκπαίδευση. Συγγνώμη, το θέμα της κατάρτιση. Είπατε ότι θα πρέπει όλοι να εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια σε ό,τι αφορά την διεκπαιρέωση των αιτήσεων για άσυλο, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ λίγα τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία έχουν πρόθεση να αποστείλουν προσωπικό προς την Ελλάδα. Η ΑΖΟ είναι μια πολύ μικρή υπηρεσία, η οποία δεν μπορεί καν να αποσπάσει πολύ προσωπικό. Δεν ξέρω και αν ε, η Επιτροπή έχει προσωπικό το οποίο θα μπορούσε να καταρτήσει για να το αποσπάσει και κοιτώντας πόσους ε, χρειαζόμαστε στη Γερμανία και ότι ακόμα δεν είμαστε σε θέση να αντιπρέσουμε τις ε, ε, αιτήσει για άσυλο και ούτε καν να τι καταχωρήσουμε. Αναρωτιέμαι, μα πώς πρέπει να συμπληρώσουμε τους αριθμούς που χρειάζονται για την Ελλάδα προκειμένου να υπάρχει μια ταχεία διαδικασία και να μπορούμε να καθορίσουμε ποιο είναι πρόσφυγα και ποιο δεν είναι. Τελευταία ερώτηση. Ότι εξακολουθούν να αρνούνται τα κράτη-μέλη να υποδεχτούν ε, πρόσφυγες. Ακόμα και αν μιλάμε για μικρούς αριθμούς. Έχετε κάποια απάντηση το τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα ή τι θα πούμε απλά ότι ε, τι να κάνουμε να τύχει σας η Ελλάδα. Θα μείνουν όλοι οι πρόσφυγες εκεί και θα δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα τα βγάλουν πέρα και να βρουν και κάποια άλλη λύση. Thank you. Um, colleagues, you may have noticed, I think Mr. didn't... Um, Συνάδελφοι, θα προσέξατε ότι δεν ε, στο θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων ο κύριος Βερβέη δεν ήταν στο πακέτο των συζητήσεων για σήμερα. Ακούει, λέει ο πρόεδρος, κάποια γλώσσα στο αυτή του. Δεν υπάρχει πάντως κάποιο πρόβλημα με την ερμηνεία. Το θέμα της απελευθέρωσης για τις θεωρήσεις θα είναι τμήματα συζητήσεις. Έχουμε ε, συναπόφαση στο θέμα αυτό. Και αν έχουμε χρόνο, αν ε, επιδείξουμε κάποια πειθαρχία. Ίσως θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε αυτό εν συντομία στο τέλος. Είναι το τμήμα του πακέτου της συμφωνίας. σε περίπτωση που δεν θεωρείτε ότι θα το συζητάμε αυτό. Ο κύριος Κέρκο από το ECR. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω πως είναι γνωστό σε όλους ότι δεν με ικανοποίησαν οι προτάσεις που αφορούν αυτή τη συμφωνία με την Τουρκία. Και πράγματι έκανα ο ίδιος κάποιες προτάσεις εκ μέρους της ομάδας μου στην Κομισιόν για το πώς θα μπορούσαν να προχωρήσουν εάν προχωρήσουν με, μια, έναν τέτοιο διακανονισμό. Ε, πολύ φοβάμαι ότι οι προτάσεις μου δεν ε, λήφθησαν υπόψη και θα ήθελα τώρα να θίξω δύο θέματα, προσπαθώντας να είμαι σύντομος. Συνεχίζω να ανησυχώ πάρα πολύ για την υλοποίηση της συμφωνίας αυτής. Ε, καταρχάς, πιστεύω πως είναι σημαντικό να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα κράτη-μέλη στηρίζουν τη συμφωνία αυτή, όχι στα λόγια, αλλά στις πράξεις. Και δεν είμαι πεπισμένος ότι αυτό συμβαίνει. Πιστεύω επίσης πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, δοθούν διευκρινήσεις για το τουρκικό σύστημα ε, ασύλου. Σύμφωνα με ε, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1951 δεν πρέπει να γίνονται διακρίσει στου πρόσφυγε με βάση την εθνικότητά του. Και πιστεύω πω ούτε και εδώ πρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτή η προσέγγιση είναι λάθο. Επίση, πιστεύω τα κονδύλια που θα ε, λάβει η Τουρκία πρέπει να ε, δοθούν με πολύ ε, μεγάλη προσοχή και με πολλές λεπτομέρειες. Πρέπει να υπάρχει μια άμεση σύνδεση των κονδυλίων με τις επιδόσεις ε, της εφαρμογής του συστήματος. Διαφορετικά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αξιολογήσουμε το πόσο αποτελεσματική θα είναι η βοήθεια. Πιστεύω επίση πως οι τουρκικές αρχές πρέπει να συμφωνήσουν σε μια ε, ανεξάρτητη αξιολόγηση από τα Ηνωμένα Έθνη και ε, αυτό να ε, αναθεωρείται κάθε τρεις ε, μήνες. Επίσης πρέπει να διεξάγεται εκτίμηση αντικτύπου κάθε έξι μήνες σε συνεργασία πάλι με τα Ηνωμένα Έθνη έτσι ώστε να δούμε εάν η ποιότητα των καταστάσεων κράτησης είναι επαρκής και αν μπορούν αυτές οι εγκαταστάσεις να φιλοξενήσουν τον ε, μεγάλο αριθμό των ανθρώπων που φιλοξενούν. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τα προγράμματα ένταξης των προσφύγων στην Τουρκία και να διασφαλίσουμε ότι αυτά θα ε, συμπεριλαμβάνουν προγράμματα εκπαίδευσης και πρόσβασης ε, στην αγορά εργασίας. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας ε, λεπτομερέστατο οδικό ε, χάρτη ε, για το πώ καταπολεμάει η Τουρκία το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και το πώ θέλουν να εφαρμόσουν τις ποινές για τους ε, διακινητές. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω πως είναι ζωτική σημασία η Τουρκία να ε, παρέχει ε, βοήθεια στην συλλογή δεκτυλικών αποτυπωμάτων των προσφύγων και να υπάρχει συνεργασία με το Eurodac. Επίσης πρέπει να υπάρχει και μια ασφαλιστική δικλίδα στο σύστημα η οποία θα ενεργοποιηθεί όταν ε, παραβιαστούν οι όροι της συμφωνίας. Και επίσης πιστεύω πως πρέπει να εμείς να μπορούμε να ε, αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο σε περίπτωση που έχουμε υπερβολικά μεγάλο αριθμό ε, ετούντων άσυλο να ε, γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μην ξεχνάτε, μπορούμε να ε, διαχειριστούμε ένα συγκεκριμένο αριθμό προσφύγων και αυτό νομίζω κάπως το ανέφερε και ε, η συνάδελφος από τους ε, σοσιαλιστές. Τα νούμερα τα οποία έχουμε δεν πιστεύω πως είναι ρεαλιστικά. Πρέπει δηλαδή να δούμε την πραγματικότητα και θα με ενδιαφέρα πάρα πολύ να ακούσω τις απαντήσεις του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των φιλελευθέρων, εντάξει δεν έχουμε και μεγάλα περιθώρια. Δεν θέλω να πω κάτι βέβαια με αυτό. Ένα μέλος έχουμε από τους φιλελεύθερους. Ναι, έφτασα μόλις τώρα. Βέβαια, κυρία Εντφέλντ, αλλά σίγουρα θα έχετε κάτι να πείτε. Δεν είστε υποχρεωμένοι, αλλά μπορείτε να λάβετε το λόγο. Θέλετε? Όχι. Περνάμε στην Google, λοιπόν. Η κυρία Ένστ έχει το λόγο. Μάλιστα. Ε, Εντάξει, δεν θα ήθελα να σκάψω το λάκκο μας η ίδια και να πω ότι βλέπω μεγάλα προβλήματα για διάφορους λόγους. Υπάρχουν όμως προβλήματα με την Τουρκία, δεν, σε, δεν γίνεται σε εμφαστό το σύμφωνο ε, της Αγενέφης για τους ε, πρόσφυγες. Δεν υπάρχουν εξηγήσεις, δεν μας έχουν εξηγήσεις ε, για το τι γίνεται με ε, τους ε, πρόσφυγες που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες στο Ιράκ. Πιστεύω πως αυτό θα έχει και συνέχεια και πρέπει να το εξετάσουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει την ε, νομική της ε, απάντηση σχετικά με το τι συμβαίνει στην Τουρκία με αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης, ε, μου είναι δύσκολο να κάνω μια γενικότερη αξιολόγηση. Γι' αυτό λοιπόν θα επικεντρωθώ σε συγκεκριμένα σημεία. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω άμεσα να δώσετε απαντήσεις στα σημαντικά ερωτήματα. Καταρχάς, ποια είναι τα κριτήρια τα οποία, ε, σύμφωνα με τα οποία αποφασίζει η Τουρκία ποιοι θα ε, προχωρήσουν στην Ευρώπη. Ποιος ε, θέτει αυτά τα κριτήρια. Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκεί έπειτα, τι γίνεται με τους πρόσφυγες που στέλνονται πίσω, ποια είναι η μοίρα τους, τι τους συμβαίνει όταν ξαναφτάνουν στην Τουρκία, παραμένουν εκεί, προχωρούν παραέξω, ποια είναι και σε αυτή την περίπτωση τα κριτήρια τα οποία αποφασίζουν τι θα γίνει. Αυτή είναι μια απόφαση που δεν πρέπει να είναι μόνο στα χέρια της Τουρκίας. Επίσης, τι θα γίνει με αυτούς τους 72.000 πρόσφυγες οι οποίοι δεν θα καλύπτονται από αυτή τη συμφωνία. Μετά από αυτούς τους 72.000 πρόσφυγες που θα ε, υποδεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα γίνει με τους υπόλοιπους. Θα δοθεί ένα τέλος, τι θα γίνει με αυτούς. Έπειτα. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η βάση στην οποία στηρίχθηκε η Ελλάδα για να αλλάξει την νομοθεσία έτσι ώστε να ε, θεωρηθούν ότι κάποιες ομάδες είναι ασφαλείς στην Τουρκία, κάποιες όχι. Πώς αποφασίστηκε αυτό. Αυτό είναι κάτι που ρώτησε και η συναδελφός μου η κυρία Ζήπελ και εγώ θα ήθελα επίσης να ε, μάθω τι συμβαίνει. Επίσης, μέχρι πότε η Ελλάδα θα ε, έχει λάβει όλη την βοήθεια που της έχει υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι κάποτε μια ώρα στη πότε θα λάβει τη βοήθεια που της έχουν υποσχεθεί. Έπειτα, τα κονδύλια που θα λάβει η Τουρκία για τους πρόσφυγες είναι ελάχιστα δισεκατομμύρια ευρώ. Εσείς όμως πώς θα διασφαλίσετε ότι τα χρήματα αυτά θα φτάσουν στην Τουρκία έτσι όπως τα έχετε προγραμματίσει. Θα διεξαχθεί κάποιος έλεγχος, θα ζητήσετε ε, αποδείξεις, θα ζητήσετε ε, εκθέσεις. Πώς δηλαδή θα γίνει αυτή η μεταφορά κονδυλίων προς την Τουρκία. Και τελευταίο ερώτημα. Πώς έχουν τα πράγματα με τα κριτήρια σχετικά με την απελευθέρωση του καθεστώτος ε, για τις ε, θεωρήσεις στην Τουρκία. Υπήρχαν κάποια προβλήματα που παραμένουν άλυτα. Τι έχει γίνει και πότε εμείς σε αυτήν εδώ την Επιτροπή πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες εξελίξεις. Thank you very much. On the aid question, uh, Mrs. McEvan, the chair of the Development Committee. Ευχαριστώ. Και μια ερώτηση από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, την κυρία Μακάβαν. Ήθελε να θέσει αυτήν την ερώτηση σε σχέση με τις ΠΚΟ και τα χρονικά όρια. Άρα λοιπόν ε, εκφράζω εδώ την ερώτηση της Επιτροπής Ανάπτυξης που έπρεπε να είναι εδώ με την Προεδρότηση. Τώρα, από το... κυρία Σαρζεντίνη από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχά, είναι κάπω παράξενο να πρέπει να συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμφωνία με την Τουρκία, όπου πολλέ σημαντικέ πτυχέ είναι σε διακυβερνητικό επίπεδο αποφασισμένε και αποφασίζονται. Εγώ θα ήθελα το Συμβούλιο εδώ να έρθει να μα εξηγήσει πώ που σκοπεύει να προχωρήσει. Και αυτό με οδηγεί στο ερώτημα πού είναι εδώ η, δημοκρατική, ο δημοκρατικός Είναι μόνο το Κοινοβούλιο της Ελλάδας. Εμείς πότε ε, παρεμβαίνουμε. Και ποιοι είναι οι ρόλοι διακριτή ανάμεσα στο Συμβούλιο και την Κομισιόν. Αυτό το ρωτώ και υπό το φως ενός άρθρου στην επικεφαλίδα, στην, μάλλον στο πρωτοσέλιδο της NRC, μια Ολλανδική Εφημερίδα, Το NRC της Τρίτης αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο της ε, Frontex της κυρία Μονκούρη ότι η ΕΑΣΟ στη Λέσβο ενημέρωσε τον κόσμο που θα έφευγε για, την Τουρκία, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Η ΕΑΖΟ όμως διατείνεται ότι αυτό δεν ισχύει, γιατί η ΕΑΖΟ δεν έχει δικαιώματα και δυνατότητες και αρμοδιότητες στα νέα κέντρα κράτησης, γιατί βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών. Θα ήθελα λοιπόν να κατανοήσω ποιος είναι ο ρόλος της ΕΑΖΟ εδώ στα κέντρα αυτά και κατά πόσον υπάρχει κάποιος ρόλος, κάποια αρμοδιότητα. Γιατί και αυτό προκαλεί πάλι μια σύγχυση μεταξύ κομισιών και διακυβερνητικών αποφάσεων σε ό,τι αφορά την κράτηση στην Ελλάδα. Σας παρακαλώ, α, πείτε μας αυτά τα, αυτά τα κέντρα ήταν ανοιχτά, αλλά τώρα είναι κέντρα κράτηση και υπάρχει έλλειψη τροφίμων. Δεν έχουν γάλα για τα βρέφη. Και αυτά συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κράτηση ατόμων χωρίς αρκετό φαγητό. Αν δεν έχουμε εξοργιστεί μέχρι τώρα, γιατί δεν έχουμε εξοργιστεί σε ό,τι αφορά τώρα την ε, έκθεση για την, για την αμνηστία, για την επιστροφή από την Τουρκία στην Συρία. Ο Επίτροπος Αβραμόπουλος θα μιλήσει στην Άγκυρα, δεν άκουσα όμως ποια ήταν τα αποτελέσματα της συζήτησης αυτής και ύστερα τα οι αριθμοί για την ε, επανατοποθέτηση για την Ελλάδα, για την ε, Ιταλία, για τη Σουηδία και έχουμε όμως πλέον μία αλλαγή των ε, αριθμών αυτών και αυτό γίνεται πλέον επανεγκατάσταση στην Τουρκία. Πώς θα γίνει η νέα κατανομή των ανθρώπων αυτών που ήρθαν στην Ελλάδα πριν στις 20 υπήρξε συμφωνία μεταξύ κρατών μελών όχι μόνο να γίνει μία εθελούσια ανακατανομή, αλλά να είναι υποχρεωτική αυτή η ανακατανομή. Μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι οποίες σταμάτησαν να λειτουργούν. Όταν τα, κέντρα αυτά έγιναν πλέον κέντρα κράτησης, ε, εξού και το πρόβλημα με τα τρόφιμα. Τι θα γίνει, η κοινωνία των πολιτών ε, απομακρύνεται. Αυτό δεν μας κουρεί τον κόδωνα του κινδύνου. Είναι η πρώτη φορά που το Κοινοβούλιο μπορεί να συζητήσει τη συμφωνία με την Τουρκία και νομίζω ότι πολλοί έχουμε ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί για τις πρακτικές ε, ε, λειτουργίες αλλά και για τα νομικά ζητήματα. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να το διευκρινίσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή πείτε μου με πάσα ειλικρίνεια ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε γιατί δεν είναι απόφαση της Κομισιόν αλλά του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Για αυτά που είπατε, υπάρχει σαφώς ένα κενό. Γιατί δεν έχουμε μαζί μας το Συμβούλιο. Αλλά σε ό,τι αφορά την γρήγορη και σημαντική εξέταση των λειτουργικών, των επιχειρησιακών ζητημάτων, σε ό,τι αφορά την κράτηση, για παράδειγμα, την έλλειψη πόρων. Είναι απίστευτα σημαντικό να υπάρξει μια πρώτη ανάλυση. Δεν υπάρχει όμως θέμα ότι υπάρχει ένα θέμα έλλειψης ε, ε, ευθύνης και το γεγονό ότι δεν έχουμε μαζί μας το Συμβούλιο. Και θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να πούμε για την ε, ευθύνη αυτή που υφίσταται. Τα μέλη τώρα λοιπόν που θέλουν να πάρουν το λόγο. Tack, herr ordförande, och eh, tack, tack till representanten från kommissionen som kom hit idag. Eh, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν που είναι σήμερα εδώ. Θα πρέπει να πω ότι οι πληροφορίες που ακούσαμε δεν με βοήθησαν να καταλάβω και να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Έχω λοιπόν ερωτήσεις. Είναι ένας κόντρα έναν όταν μιλάμε για αυτή τη συμφωνία. Μα δεν είχε όμως προβλεφθεί να έχουμε επιστροφή ενός πρόσφυγα σε ανάλλαγμα ενός άλλου. Δεν ισχύει αυτό. Και έπειτα να θυμίσω ότι έχουν φτάσει 202 άνθρωποι από την Ελλάδα στην Τουρκία. <clears throat> σε ένα σκάφος και από όλους αυτούς μόνο δύο ήταν Σύριοι. Ενώ στην ίδια περίοδο κάποιοι μετεγκαταστάθηκαν. Πώς λειτουργεί τελικά αυτή η συμφωνία. Υπήρχαν ε, Αυγανοί, Πακιστανοί, Ιρακινοί, μόνο δύο Σύριοι. Πώς υπολογίζονται ακριβώς αυτή η ανταλλαγή λοιπόν ένας κόντρα έναν. Έπειτα, οι ποσοστώσεις. Όντως, Φτάσανε, λέει, 172 άνθρωποι. Ε, μάλλον, εμείς, ε, ε, μάλλον η Τουρκία πω, τι θα κάνει όταν φτάσει σε αυτή την ποσόστοση. Θα πάψουμε να τους στέλνουμε. Τα κράτη-μέλη τι κάνουν. Ή θα διαπραγματευτούμε νέα ποσόστοση. Γιατί, ας πούμε, η Σουηδία είναι σε αυτή τη φάση. Δεν έχουμε πια χώρο. Και αυτό για την αναγκαστική υποχρεωτική με την κατάσταση δεν περνάει, δεν αρέσει. Στη συνέχεια, χρηματοδότηση. Ξέρουμε ποιος θα πληρώσει πόσα εκατομμύρια, πόσα θα δώσει η ε, Σουηδία για παράδειγμα. Ξέρετε ακριβώς τα ποσά για κάθε χώρα. Ευχαριστώ. Κύριε εγώ έχω, έχει μάλλον ήδη τεθεί ερώτηση, αλλά επιμένω γιατί όταν ακούω πώς εξηγεί την εφαρμογή αυτού του σχεδίου η Κομισιόν, έχω την εντύπωση ότι στην ουσία φτιάχνουμε ένα μηχάνημα, ένα τέρας, ένα τερατώδες πράγμα ε, και πάντως αυτή είναι η αίσθηση που έχουμε. Είναι μια αίσθηση που είναι κοινή για ορισμένες ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς, γιατί Ορισμένες ε, υπηρεσίες ε, είναι παράξενες. Ας πούμε, πώς αντικαθιστούμε, πώς καλύπτουμε αυτή την απουσία, αυτή την απόσυρση ορισμένων υπηρεσιών επιτόπου. Είπατε ότι είναι ότι λιγότεροι αυτοί που περνούν, λιγότεροι άρα νεκροί, αυτό που είναι λογικό. Αλλά δεν μας είπατε ότι από ό,τι φαίνεται παράλληλα υπάρχουν πολύ περισσότερα αιτήματα ασύλου. Θέλω να έχω την εκτίμησή σας ε, για το κατά πόσο οι ελληνικές αρχές είναι σε θέση να εξετάσουν αυτά τα αιτήματα και τα ενδεχόμενες προσφυγές που μπορεί να γίνουν, γιατί οι διαδικασίες, όπως είπαν ε, κάποιοι συνάδελφοι, δεν είναι ακριβώς ε, οι ίδιες παντού. Το δεύτερον, ε, η ευαισθησία της νομικής βάσης αυτής της ε, συμφωνίας, όπως και ο ε, δημοκρατικός έλεγχος που απουσιάζει από όλα αυτά, πώς όλα αυτά συζητήθηκαν και λύθηκαν από το Συμβούλιο και έπειτα για να, χωρίς να μιλήσω πολύ για τα δις, ε, ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το κόστος όλων αυτών των ε, δραστηριοτήτων, όχι μόνο τα τρία δις επιμένω, αλλά και τον τρόπο χρηματοδότησης του επιπλέον κόστους ε, αυτών, για αυτές τις δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Η κυρία Σπινέλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύμφωνα με μια νομική ανάλυση της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ στις 10 Μαρτίου, η μεταφορά των ετούντων άσυλο από μια ευρωπαϊκή χώρα σε μια εξωευρωπαϊκή χώρα θα πρέπει να σέβεται μια ολόκληρη σειρά ελάχιστων εγγυήσεων. Είναι καταρχάς σημαντικό το κράτος υποδοχής να αναλαμβάνει την ευθύνη να παρέχει πρόσβαση στους ετούντες άσυλο σε ένα ε, σύστημα ασύλου ε, υποδεχόμενοι και ε, καταγράφοντας τα αιτήματα προστασίας. Το κράτος υποδοχής θα πρέπει να αξιολογεί τα αιτήματα ασύλου επί της ουσίας ε, σύμφωνα με μια ισότιμη διαδικασία. Το κράτος υποδοχής πρέπει να, να προστατεύει τους ετούντες σε άσυλο από την απόθεση, όπως προβλέπεται εδώ και 65 χρόνια από τη Σύμβαση της Γενέβης. Οι πρόσφυγες δεν πρέπει να έπαν επιστρέφονται σε περιοχές που σοβούν πολεμικές σειράξεις και οι σε άσυλο, αν, αν αναγνωριστεί το, το καθεστώς πρόσφυγα, θα πρέπει το κράτος υποδοχής να εξασφαλίζει την προστασία σύμφωνα με εγγυήσει και διεθνείς προδιαγραφές. Αυτή τη στιγμή καμιά από αυτές τις εγγυήσει δεν τηρείται από την Τουρκία. Γι' αυτό και ζητώ να ανακληθεί αυτή η συμφωνία πριν να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπου θα καταργήσουν αυτή την τροπή. Το ζητούν μαζί με μένα και την ομάδα μου 90 ευρωπαϊκές ενώσεις που ασχολούνται με τους πρόσφυγες. Η Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα. Και μια ερώτηση επί της ουσίας κύριε Βερβέ. Μην επαναπαύεστε τόσο με αυτή την συμφωνία που κάνατε, ούτε να χαίρεστε, γιατί όταν μιλάτε για νούμερα για τις επιστροφές σας, παρακαλώ να αναφέρετε τις εκατοντάδες πρόσφυγες που έχει διώξει η Τουρκία προς την Συρία. Είναι χιλιάδες. Εδώ και 7-8 μήνες γίνεται αυτή η δουλειά. Και παιδιά που τα στέλνουν πίσω στη Συρία χωρίς το καν γονείς, τους γονείς τους, μόνο τους. Και σας ζητώ να μην κρύβετε τα όσα συμβαίνουν στα κέντρα κράτησης στην Ελλάδα. Η κατάσταση ήδη έχει περιγραφεί τέλεια από τη συνάδελφο Σαρτζεντίνη. Μην κρύβετε το ότι δεν λειτουργεί σε αυτή την συμφωνία. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την εισήγησή σας που όντως αφήνει πολλά εκκρεμή ερωτήματα, πολλά εκ των οποίων ετέθησαν. Θέλω να προσθέσω μπορείτε να διευκρινίσετε τις αλλαγές στην νομοθεσία στις οποίες προέβη η Τουρκία σε σχέση με την προστασία των προσφύγων. Ο Πρωθυπουργό Νταβούτογλου είπε ότι η Τουρκία δεν θα κυρώσει τη συμφωνία της Γενέβης με όλα τα ε, πρωτόκολλα κτλ. Και το δικαίωμα στην εργασία ήταν μια από τις λεπτομέρειες που υποτίθεται έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί. Πείτε μας λοιπόν τι συμβαίνει. Επίσης είπατε ότι η Τουρκία θα θεωρηθεί ε, ασφαλή για, ασφαλής για ορισμένες ομάδες. Μα ποιες ομάδες και γιατί ομάδες, γιατί από όσο ξέρω η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι σαφής για την ατομική αξιολόγηση. Εσείς υπο, λέτε ότι θα υπάρξει αλλαγή ώστε τα ατομικά ε, αιτήματα για άσυλο ε, δεν θα κρίνονται ατομικά, αλλά θα σχετίζονται με ομάδες εθνικοτήτων. Μετά υπήρξε ανακοινωθέν από την Κομισιόν ότι οι πρόσφυγες που καταφτάνουν μετά από τις 20 Μαρτίου αλλά που αλλά που εκτιμάται ότι δεν είναι ασφαλή στην Τουρκία και φτάνουν στην Ελλάδα και ζητούν άσυλο, δεν θα είναι επιλέξιμη για επανεγκατάσταση. Γιατί δεν υπάρχει ε, χρονική προθεσμία στην απόφαση για επανεγκατάσταση, γιατί η Κομισιόν ε, έφτιαξε άλλη μία προθεσμία. Εφόσον δεν μπορεί να το κάνει, δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση. Στη συνέχεια είπατε ότι σας ανησυχεί η κατάσταση που επικρατεί στα, ε, στα τόπεδα κράτησης. Ναι, αλλά και τι κάνετε που ανησυχείτε. Τι βοήθεια έχει δοθεί, χρήματα, πόσα, πότε, με τι τρόπο. Τα δίνετε όταν ε, ε, έχουν στείλει το λογαριασμό. Θέλουμε να τα έχουμε και γραπτός αυτά αν γίνεται. Και για το γεγονός ότι έρχονται λιγότεροι από, την, ε, από το Αιγαίο, θα ξέρετε βέβαια ότι τώρα οι διακινητές προσφέρουν και την πολύ μακρύτερο, μακρύτερο δρόμο από μέσω της Ιταλίας ε, όπου είναι πολύ πιο επικίνδυνος ο δρόμος γιατί είναι πολύ περισσότερα χιλιόμετρα και δεν είμαι βέβαιη ότι θα πεθάνουν λιγότεροι. Ε, θέλω λοιπόν να απαντήσεις. Αρκετοί συνάδελφοι είπαν ότι θέλουν να απαντήσεις. Αυτό καθιστά σαφές ότι δεν ε, έχουμε πια διαρκώς απαντήσεις από την Κομισιό, αλλά θα ήταν ωραία αν εσείς ήσασταν η εξαίρεση στον κανόνα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ράντεφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τους τελευταίους μήνες έχει καταστεί σαφές ότι αυτή η μεταναστευτική κρίση σημαίνει πως πρέπει να συνεργαστούμε. Όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τις γειτονικές μας χώρες, ιδιαίτερα με την Τουρκία. Η συμφωνία με την Τουρκία μπορεί να μην είναι η χρυσή λύση, όμως σίγουρα θα χαμηλώσει την ε, πίεση που δέχεται η Ευρώπη. Και οι Σύριοι πρόσφυγες θα μπορούν επιτέλους ε, να απολαμβάνουν διεθνούς προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσοι έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ε, να έχουν κάποια νομική βάση θα ξέρουν ότι δεν θα μπορούν να παραμείνουν. Σίγουρα βέβαια η αστυνομία πρέπει να συνεργάζεται και, με, και η βουλγαρική με την τουρκική και σίγουρα η Ελλάδα θα πρέπει να καταπολεμήσει τη, τα δίκτυα διακινητών. Η Βουλγαρία, από την άλλη, θα πρέπει να προσπαθήσει να σταματήσει ε, αυτούς τους ε, διακινητές κλείνοντας ε, τις ε, οδούς που χρησιμοποιούν. Αυτό που χρειάζεται επίσης είναι να ενισχυθεί η ασφάλεια στα συνορα βουλγαρια Βουλγαρίας-Τουρκίας, διότι διαφορετικά πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα βρουν καινούριο ε, δρόμο οι διακινητέ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να πάρετε το λόγο. Κύριε Κύρκο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα πρέπει ε, να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, να μην αφήσουμε τους πρόσφυγες να θαλασσοπνίγονται και να τους φέρνουμε με ασφάλεια στην Ευρώπη. Άκουσα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ε, απάντησή σας στον Πρόεδρο για τους ε, αξιωματούχους που θα έρθουν στην Ελλάδα και που ήδη έχουν φτάσει. Έχετε εσείς κάποια παραπάνω πληροφορία για το πότε επιτέλους θα έρθουν αυτοί οι υπάλληλοι που θα βοηθήσουν ε, τις ελληνικές αρχές στην επεξεργασία των ε, ετοιμάτων ασύλου. Είδαμε πολλές φορές πολλές εμίκιο να αποχωρούν από τις εγκαταστάσεις κράτησης και να μην έχουν λοιπόν οι πρόσφυγες φαγητό, να μην έχουν στέγη, και ιατρική ε, περίθαλψη. Αυτή η συμφωνία λοιπόν ε, δεν έχει υλοποιηθεί και δεν φταίμε εμεί ε, γι' αυτό. Όπως είπε και η κυρία Βόζεμπεργκ, αυτή τη στιγμή όλοι οι άνθρωποι που έρχονται στην Ελλάδα ζητούν να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες. Εμείς δεν έχουμε τα μέσα να διαχειριστούμε τον όγκο αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα ήθελα να ε, σας ε, κάνω το εξή ερώτημα. Πόσο καιρό νομίζετε πως θα αντέξουν αυτά τα κέντρα υποδοχής χωρίς να ε, διαλυθούν τα πάντα. Δεν έχουμε την διοικητική δυνατότητα να διαχειριστούμε όλα αυτά τα αιτήματα ασύλου και να ξέρετε υπάρχουν κάποιες βάρκες που ακόμα φτάνουν ε, στην Ελλάδα και τα hot spot δεν ε, μπορούν να υποδεχτούν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθούμε κάθε μέρα να βρούμε λύση στα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά είναι πάρα πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν και πολύ ωραία παρέμβαση για να ολοκληρώσουμε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι ερωτήσεις και πιστεύω πως προτού τις απαντήσετε θα πρέπει να ε, διασφαλίσετε ε, την μεταφορά αυτών των προβληματισμών και των ερωτήσεών μας στους ε, συνεργάτες σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όπως είπε και η κυρία Σαρτζεντίνη, δεν σας ζητούμε να λογοδοτήσετε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τουλάχιστον μας δώσετε λεπτομέρειες, διότι στις λεπτομέρειες βρίσκονται πάρα ε, πολλά σημαντικά στοιχεία. Σίγουρα η πίεση που σας ασκείται είναι μεγάλη, όμως αυτό είναι και ένα μέρος της δουλειάς σας. Δεν μπορώ λοιπόν να δείξω κατανόηση αν μου πείτε ότι εντάξει έχω μεγάλες πιέσεις. Το επιλέξατε. Σας παρακαλώ λοιπόν να απαντήσετε στις ερωτήσεις των μελών. Έχουμε αρκετό ε, χρόνο που έχουμε κρατήσει για εσάς. Γι' αυτό λοιπόν Έχετε το λόγο και προσπαθήστε να απαντήσετε όσο το δυνατόν καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Για να είμαι ειλικρινής, ε, δεν περίμενα να δείξετε κατανόηση στο πρόσωπό μου. Όπως είπατε και εσείς, η δουλειά μου συνεπάγεται μεγάλη πίεση. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια και για όλες τις ερωτήσεις που κάνατε. Αναφέρθηκαν σοβαροί προβληματισμοί από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να είστε σίγουροι πως θα τους μεταφέρω στους συνεργάτες μου. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να δώσω κατάλληλες απαντήσεις σε αυτούς τους προβληματισμούς. Σίγουρα ίσως να μην καταφέρω να απαντήσω σε όλες ε, τις ερωτήσεις, όμως σας διαβεβαιώ ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι είναι ανθρώπινα δυνατό έτσι ώστε όχι μόνο να ε, έχουμε μια επιτυχημένη συμφωνία, αλλά και μια συμφωνία επιτυχημένη έτσι ακριβώς όπως το ε, επιθυμούμε και έτσι όπως πρέπει να είναι. Πρέπει να έχουμε λοιπόν μια συμφωνία που θα συμφωνεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτά ως ε, αρχή. Τώρα, Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω, διότι είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποια κενά στην πληροφόρηση και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αρχίζω λοιπόν με αυτό. Ακούστηκε ότι το 5% των ε, ανθρώπων που φτάνουν ε, στην Ευρώπη ζητούν άσυλο. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Από όσο ξέρω, 4.261 άνθρωποι ε, ζήτησαν άσυλο. Σίγουρα είναι μεγάλος ο αριθμός, όμως δεν είναι το 95% των όσων φτάνουν. Επίσης, δεν πρέπει να βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα προτού δούμε ε, τις ε, ατομικές ε, αιτήσει ασύλου όσων βρίσκονται στην Ελλάδα. Πιστεύω μάλιστα πως ένας μεγάλος αριθμός αυτών των ανθρώπων θα επιστραφεί. Και να πω ότι σίγουρα η αξιολόγηση πρέπει να γίνει για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Θα είμαι σαφής λοιπόν. Οι αλλαγές που έχουν γίνει στην Τουρκία για τους Σύρους και να σας υπενθυμίσω εδώ ότι η Τουρκία φιλοξενεί πάρα πολλούς Σύρους, δείχνει μια ξεκάθαρη δέσμευση, η οποία έχει μεταφερθεί στην ε, τουρκική νομοθεσία. Οι Σύροι επιστρέφ, που θα επιστραφούν από τα νησιά στην Τουρκία θα λάβουν αυτό το καθεστώς προσωρινής προστασίας, το οποίο είναι απόλυτα συμβατό με το διεθνές δίκαιο και με όλες τις σχετικές συμβάσεις. Επίσης, είναι επίσης σαφές ότι πριν ακόμα από τη συμφωνία βασισμένη στις διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία ήταν ε, δυνατό να επιστραφούν αυτό που ονομάζουμε οικονομική μετανάστες, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα διεθνούς προστασίας. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο μέρος ε, όσων φτάνουν στην Ελλάδα αυτοί οι οικονομικοί μετανάστες και είμαι σίγουρος πως αυτό θα συνεχιστεί να παραμένει υψηλό. Επίσης, ε, διατυπώθηκαν πολλές ερωτήσεις σχετικά με την ε, μετακατάσταση. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και συγκεκριμένες δεσμεύσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να κάνει τα κρατημέλη να τηρήσουν αυτές τις δεσμεύσεις τους. Τώρα γιατί είπα ότι αυτό αφορά όσους έφτασαν πριν τις 20 του μήνα, ε, διότι πριν δεν είχε γίνει κάποια ε, αλλαγή του νομικού καθεστώτος, αλλά και επειδή όσοι φτάνουν μετά τις 20 θα επιστραφούν στην Τουρκία, εκτός εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ε, συνθήκες που θα επικρατούν και αυτό θα αποφασιστεί βάσει ατομικής αξιολόγησης. Τώρα, σε σχέση με το αν υπάρχουν επαρκείς δεσμεύσεις για μετεγκατάσταση προσφύγων. να σας πω ότι προς το παρόν 55.000 άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα. Δεν είναι όλοι αυτοί επιλέξιμοι για τα προγράμματα μεταγκατάστασης. Και πιστεύω πως από του ανθρώπου που βρίσκονται στην Ελλάδα θα μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα μετακατάστασης 66.000. Αυτό είναι ένα νούμερο που ε, το λέω από μνήμης δεν... Μην το θεωρήσετε ακριβές. Βρίσκεται όμως ακόμα να εξελίξει αυτή η συζήτηση. Τώρα, σχετικά με το αν υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση. Είναι πολύ καλή ερώτηση. Και μπορώ να σας πω ότι για μένα καμία λύση δεν είναι τέλεια. Και πρέπει να αποδεχτούμε το ότι η κατάσταση αυτή ε, δεν είναι εύκολη. Είναι χαοτικά τα πράγματα, άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, τίποτα δεν είναι εύκολο, δεν μπορεί να υπάρξει εύκολη και καλή λύση. Πιστεύω όμως πως αυτή η συμφωνία που έχουμε τώρα είναι αρκετά περιεκτική και μπορώ να δεχτώ την κριτική και τις διαφορετικές απόψεις πολλών, όμως πιστεύω ότι από αυτή την κριτική και, τις, ε, και τους προβληματισμούς ε, Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να επιλύσουμε. Τώρα, ας ε, απαντήσω σε κάποια άλλα ερωτήματα. Πώς θα αξιολογηθεί η κατάσταση κατά ομάδες ή ε, κατά άτομο. Σας ε, το είπα, ατομική αξιολόγηση παραμένει ως έχει. Είναι, είναι ο μόνος τρόπος για να γίνει κάτι ε, νόμιμα. Εγώ προσωπικά δεν επεξεργάζομαι τη ασύλου, όμως σας διαβεβαιώ ότι θα γίνεται ατομική αξιολόγηση των ε, ετοιμάτων. Έτσι έχει το σύστημα που θα εφαρμοστεί. Επίσης, αναφέρθηκαν ανησυχίες για το τι θα γίνει με ε, ανθρώπους άλλης εθνικότητας. Και εδώ επαναλαμβάνω ότι οι αξιολογήσεις θα είναι ατομικέ. Σίγουρα βέβαια είναι αναμενόμενο ότι οι οικονομικοί μετανάστες δεν θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους πρόσφυγες. Αυτό βέβαια και πάλι ε, θα αποφασίζεται μετά από ατομική αξιολόγηση. Επίσης, όπως ανέφερα, οι συζητήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και επίσης να επαναλάβω ότι θα ε, επιστρέφουν άτομα με νόμιμο τρόπο. Τώρα, όπως είπα και πριν, η ΕΑΣΟ θα αυξήσει το προσωπικό της. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει να υπάρχει προθυμία από τα κράτη-μέλη για να στείλουν τους εμπειρογνώμονες, να στείλουν αρκετό προσωπικό και αυτό θα γίνει σταδιακά, όμως θα αυξηθεί σταδιακά το προσωπικό και οι δυνατότητέ μας. Μάρτιν, μία ερώτηση. Ξέρεις, το θέμα αυτό το σε μία νύχτα. Είπατε ότι έχουμε 30 εκπαιδευμένα άτομα θα πρέπει να περάσουν από τη σχετική κατάρτιση. Μιλάτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ υπάρχουν πολλοί εμπειρογνώμονες με υψηλό βαθμό κατάρτισης. Φαντάζομαι ότι πολλοί θα είναι οι εθελοντές οι οποίοι θα ήθελαν να μεταβούν εκεί επί τόπου για να αξιολογήσουν τις αιτήσει αυτές. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι στο μυαλό πολλών συναδέλφων, γιατί έχει εκφραστεί σε διάφορες συναντήσεις. Θα ήθελα να εκφράσω κάποιες από τις πιο βαθιές ανησυχίε μας. Βλέπουμε ότι υπάρχουν εκεί λοιπόν 30 εκπαιδευμένα άτομα και μας λέτε ότι παίρνει πολύ χρόνο η εκπαίδευση τι εκπαίδευση για, να είναι κανείς στην Ελλάδα σε συνθήκες αυτές είναι υποκράτηση, θα υπάρχουν και άτομα από άλλα κράτη-μέλη, υπάρχουν αξιωματούχοι. Ο διάολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και πιστεύω ότι θα μπορούσε να καταρρεύσει όλο το σύστημα. Αν έχουμε 30 άτομα αντί για 400, είναι μεγάλο επιχειρησιακό το ζήτημα αυτό. προδιαγραφές, τι προϋποθέσεις υπάρχουν για την εκπαίδευση που καθυστερούν τη διαδικασία. Γιατί δεν μπορεί να γίνει ε, ατομική εξέταση των αιτήσεων με τον τρόπο αυτό. Να σας εξηγήσω. Να σας εξηγήσω. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση δεν διαρκεί πολύ. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια κοινή κατανόηση του πώς ε, αξιολογούνται οι αιτήσει. Αυτή την εβδομάδα, για παράδειγμα, για την πρώτη ομάδα έγινε μια εκπαίδευση μία μισή ημέρας. Δεν είναι τεράστια τα πακέτα εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά να μην είναι απροετοίμαστο ο κόσμος. Όσοι έχουν σε κάποια διευθυντική θέση στο παρελθόν θα ξέρουν ότι υπάρχουν και όρια στο πόσο γρήγορα μπορεί να κινηθεί κανείς. Να σας διαβεβαιώσω ότι ε, προσπαθούμε να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά θα πρέπει και ο κόσμος να απορροφηθεί από το σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν δεν μιλάω για χρόνια και μήνες. Γρήγορα θα αναπτυχθεί το σύστημα. Αλλά θα χρειαστεί μια βαθμία προσέγγιση και θεωρώ ότι αυτός είναι ο υπεύθυνο τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος. Γιατί μόνο με μια οργάνωση που λειτουργεί μπορεί να πετύχει κανείς αποτελέσματα. Αυτό είναι απλή διευθυντική λογική. Ο Πρόεδρος. Για τα λειτουργικά αυτά ζητήματα νομίζω ότι τρία, α, τρεις βουλευτές ήθελαν να ξαναπάρουν το λόγο. Ε, έχετε αντίρρηση? Α, εν συντομία όμως, συνάδελφοι. Πολύ, πολύ σύντομα η κυρία Ένστ Γκυγιόμ και Σίπελ. Σας παρακαλώ όμως πολύ σύντομα να θέσετε τις διπλωματικές ερωτήσεις σας. Η κυρία Ένστ, παρακαλώ, ερώτηση. Ως τώρα, θεωρούσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν εταίρος μας, με τον οποίο μπορούμε να συνομιλούμε ανοιχτά. Είχαμε τις δυσκολίες μας στο παρελθόν, δεν λέω, αλλά μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά. Σα παρακαλέσαμε συγκεκριμένα να απαντήσετε, με συγκεκριμένε απαντήσεις, σε συγκεκριμένε ερωτήσεις. Δεν απαντήσατε ούτε μία από τις επτά ερωτήσεις που έχω θέσει. Δεν περιμένω ότι θα είσαστε σε θέση να μιλήσετε και να απαντήσετε σε όλε τι ερωτήσει, αλλά δεν είναι δυνατόν να κινούμαστε έτσι, Σκανδαλώδε. Και το τονίζω αυτό. Δεν είμαστε... Ε, έτσι μια κοινότητα της πλάκας, είμαστε κοινοβούλιο. Έχουμε δικαίωμα για απάντηση και ίσως αυτό δεν έφερε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους. Ε, ο κύριος Βέρνερ έχει ακόμα χρόνο στη διάθεσή του για να απαντήσει, λέει ο πρόεδρος. Νόμιζα ότι θέλετε να κάνετε μια επιπρόσθετη ερώτηση, κυρία Ένς. Η κυρία Γεγιόμ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να μας απαντήσετε. Όταν μιλήσατε για τον αριθμό των ατόμων όμω 30, 32, που θα πρέπει να εκπαιδευτούν και να περάσουν μια εκπαίδευση μια μια μισή ημέρα. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αξιωματούχοι από άλλα κράτη-μέλη Ποιοι είναι λοιπόν. Και ανάλογα με το από πού προέρχονται, πιστεύετε ότι αρκεί μια, μια μισή ημέρα για να τους καταρτήσετε. Ποιοι είναι, εν πάση περιπτώσει, ο Και η κυρία Σίπελ, σας παρακαλώ και εσείς πάρα πολύ σύντομα για να ζητώσουμε το λόγο στον κύριο Βεργέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να επανέλθω στο ερώτημα που είχα θέσει. Ποιος προστατεύεται στην Τουρκία, είπατε στην απάντησή σας, οι Σύριοι. Και κατά τα άλλα υπάρχουν και οικονομικοί μετανάστες. Αλλά εγώ ποτέ δεν χρησιμοποιώ τον όρο του οικονομικού μετανάστε, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από την ένδυα. Τι γίνεται με τους Ιρακινούς, τους Αφγανούς, τους Κούρδους, οι οποίοι από όσο γνωρίζω δεν, έχουν, δεν λαμβάνουν το καθεστώς του πρόσφυγα στην Τουρκία. Και ρωτώ λοιπόν πώς μπορεί αυτό να συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο να ε, επιστρέφουμε άτομα σε χώρες όπου δεν υπάρχει ασφάλεια και δεν μπορούν να προστατευτούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ε, δεν έχουν καταλήξει τελικά σε μια αμφιλεγόμενη συμφωνία Ακόμα και αν συμφωνούσαμε τη συμφωνία αυτή, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί. Καταστροφικό. Μία ερώτηση λοιπόν σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Ελπίζω τα πρότυπα τα οποία που έχουν να κάνουν με την απελευθέρωση των θεωρήσεων να μην υπονομευθούν. Εκτός μικροφώνου ο Α, μάλιστα. Συγγνώμη που σας διάκοψα. Έχετε το λόγο και πάλι για να απαντήσετε. Ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί της ΕΑΖΟ, ήταν η ερώτηση της κυρία Γκίγιον. Αναλυτέ, εμπειρογνώμονε που έχουν συνηθίσει και κάνουν τέτοιου είδου δουλειά. Ε, η εκπαίδευση δεν έχει να κάνει με την εκμάθηση της δουλειά. Απλά θα πρέπει να υπάρχει μια συνοχή, μια συνέπεια στη λήψη αποφάσεων. Η τελική απόφαση δε λαμβάνεται υπό το ελληνικό δίκαιο, από τους Έλληνες ε, ηθήνοντες. Γίνεται μια προετοιμασία των αποφάσεων, αν θέλετε, προκειμένου να υπάρχει ε, καλύτερη ανάπτυξη των ικανοτήτων. Αλλά τελικά είναι ελληνική η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Αφετέρου η νομιμότητα ενός συστήματος μπορεί να αξιολογηθεί μόνο εκ των υστέρων. Μετά τη λήψη αποφάσεων, το έχω επαναλάβει αυτό συχνά, ότι οι αποφάσεις αυτές θα βασίζονται σε μία εξατομικευμένη λήψη αποφάσεων. Να συνεχίσω λοιπόν με τις υπόλοιπες ερωτήσεις. σημειώνω τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για τις άλλες εθνικότητες. Όπως διευκρινίσα, βρισκόμαστε σε φάση συζήτησης για τα ζητήματα αυτά. Notes Σημείωσα. τα σχόλια και τις συστάσεις. σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την εποπτεία για τη χρηματοδότηση που χορηγείται. Να σας πω ότι μιας και μιλάμε για την ταπάνη ενός μεγάλου τμήματος του προϋπολογισμού, ισχύουν οι συνήθεις κανόνες σε ό,τι αφορά και τα θέματα εποπτείας. Τι κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν για την επανεγκατάσταση, ρωτήσατε. Θα βασιστούμε σε μεγάλο βαθμό στα κριτήρια ε, του ΟΗΕ για το πώς, κατά πόσο πρόκειται για ευάλωτα άτομα. Τι θα γίνει αν ξεπερθεί το όριο των 73.000. 72.000. Υπάρχει τώρα μια συμφωνία για τις 72.000. Δεν μπορώ να εικάσω και να σας πω τι θα γίνει μετά Και να προδικάσω τι θα συμβεί μετά τις 72.000. Δεν είναι στις αρμοδιότητές μου. ερώτηση επίση ακούσαμε για το τροποποιείται και η νομοθεσία στην Ελλάδα. Προσπάθησα να εξηγήσω στο σημείο αυτό ότι η Ελλάδα έχει συμπεριλάβει στα, στην νομοθεσία της κριτήρια για να καθορίζεται το κατά πόσον μία χώρα, μια τρίτη χώρα είναι ασφαλής ή όχι, ή αν αποτελεί χώρα ασύλου. Και ανάλογα ενδεχομένως αυτό να αποτελέσει κριτήριο για τη μη παραδεκτότητα του αιτήματο της αίτησης. Και ανάλογα ισχύουν και οι δικαστικές ε, Σχετικέ ε, συνέπειε. Δεν είμαι ε, ειδήμων, αλλά θεωρώ ότι αυτέ είναι οι βασικέ αλλαγέ. Για τις ΜΚΟ που σταμάτησαν τις εργασίες τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο για μένα να σχολιάσω το γεγονός αυτό. Κάθε μη κυβερνητική οργάνωση, κάθε οργάνωση λαμβάνει τις αποφάσεις της. Εγώ δεν μπορώ παρά να τη σεβαστώ. Κάποιες ΜΚΟ πολύ απλά έχουν καταστατικό που προβλέπει ότι δεν μπορούν να δραστηριοποιούνται σε κλειστά κέντρα. Αυτό δεν μπορώ παρά να το δεχτώ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε και το κάναμε μάλιστα, είναι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση η οποία προκύπτει στη συνέχεια. Παρέχαμε κατεπίγουσα βοήθεια 30 εκατομμύρια, εάν σωστά ενθυμούμε, για τα τρόφιμα, για τον καθαρισμό, για ιατρικές ε, υπηρεσίες, για τα βασικά και στοιχειώδη. Και αυτό λειτουργεί, έξω όσο γνωρίζω. Αλλά προφανώς, και εδώ δεν θέλω να κρύψω το οτιδήποτε, προφανώς η κατάσταση στα κέντρα αυτά, τα κλειστά αυτά κέντρα δεν είναι ιδανική, γιατί υπάρχει υπερβολικά μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού. Θα συνεχίσουμε όμως τις εργασίες μας προς την κατεύθυνση αυτή. Και εγώ ασφαλώς και θα καλωσόριζα την επιστροφή των ΜΚΙΟ και κάποιες από αυτές έχουν όντως ήδη επιστρέψει. Μία άλλη ερώτηση για το ύψος της χρηματοδότησης. για τα χρήματα για την Τουρκία. Υπολογίσαμε ότι έχουμε 270 εκατομμύρια για την ε, εφαρμογή για τον επόμενο χρονικό διάστημα. Θα σταματήσω στο σημείο αυτό και ζητώ συγγνώμη για ενδεχόμενες αναπάντητες ερωτήσεις. Αυτό τώρα επαφείται στον Πρόεδρο. Okay, thank you very much for, for those answers. So, colleague... Σας ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις αυτές. Συνάδελφοι, Είναι λίγο δύσκολο να κάνω μία σύνοψη, αλλά καταρχάς θα θέλαμε, κύριε Βερβέη, καταρχάς να επιστρέψετε εδώ πέρα στην Επιτροπή μας για να μας ε, αναφέρετε για τα επιχειρησιακά ζητήματα. Ήταν δύσκολη, αν θέλετε, αυτή η συνάντηση, αλλά αναγκαστικά είναι δύσκολη, γιατί πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις που πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι ανησυχίε προέρχονται από όλο το πολιτικό φάσμα. Είναι βαθιέ ανησυχίε για τα νομικά ζητήματα, τα επιχειρησιακά ζητήματα, τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κυρία Σαρτζεντίνη έθιξε το θέμα του διακυβερνητικού χαρακτήρα. Φυσικά υπάρχει έλλειμμα εδώ σήμερα. Για να σας πω με πάσα ειλικρίνεια, δεν έχω δει θέμα όπου ενδεχόμενα επιχειρησιακά ελλείμματα να απειλούν την καταστροφή όλου του συστήματος και να επαπειλούν με ξέσπασμα ανθρωπιστικής ε, κρίσης. Ακούσατε λοιπόν τι ανησυχίε που εκφράστηκαν εδώ σήμερα. Σα παρακαλώ να παραμείνετε σε επαφή μαζί μα και να μα ενημερώνετε για τι εξελίξει και θα θέλαμε πραγματικά να σα ξαναδούμε. Σας ευχαριστώ και πάλι, συνάδελφοι, για την πειθαρχία που επιδείξατε σήμερα και για τις ερωτήσει που θέσατε. Colleagues, we have votes at 10.45. Συνάδελφοι, στις 10 και 45 είναι η ψηφοφορία. Μην απομακρυνθείτε. Για να ξεκινήσουμε στις 10 και 45. Because the votes are about to begin, but you don't seem to be... Λοιπόν, συνάδελφοι, ε, θα αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Καθίστε παρακαλώ. Colleagues, it's all electronic, so have your voting cards ready. Ε, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε, οπότε παρακαλώ να έχετε τις κάρτες σας. Αν κάποιος δεν έχει την κάρτα του, ας μας το πει. Εάν δεν το έχετε, δεν έχετε, θα, θα δούμε τι κάνουμε. καθώς κάθεστε όλοι, να ανακοινώσω ότι η κυρία Κοράτσα Μπέλτ έχει καλέσει μια ομάδα Σουηδών φοιτητών. Ε, καλωσορίσατε. Ήρθαν στην Επιτροπή μας να δουν πώς δουλεύουμε. Okay, is everyone ready? Είστε όλοι έτοιμοι? Θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία για την εφαρμογή τις οδηγίες ε, για την πρόληψη και την καταπολόμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων με γνώμονα την ισότητα των φύλων. Μάλλον είναι η συγγήτρια. Ε, Μάλλον Μπιόρκ θέλετε το λόγο. Όχι, πάμε στη εμπιστοφορία κατευθείαν. Και ξεκινάμε με την τροπολογία 33. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Compromise 3, the vote is open. Συμβαστική 3, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37, Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Πρώτο τμήμα. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Άρχεται. Διάλειμμα για ένα λεπτό. Είμαστε στη συμβαστική 5. Συμβαστική 5 άρχεται τώρα. Closed. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 51. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53. 53. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 54. Άρχεται. Closed. Rejected. Amendment... Απορρίπτεται. 55. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. 58. Άρχεται. Τέλος. 59. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. 61. Πρώτο τμήμα. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. 64. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. 65. Άρχεται. Τέλος, εγκρίνεται. Τροπολογία 66. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. 67. Άρχεται. The vote is closed. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 68. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 69. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6, πρώτο τμήμα, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία ε, συμβιβαστική, συγγνώμη, 6, δεύτερο τμήμα, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. 77. Τέλος. That's carried. Εγκρίνεται. 78 άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 80, πρώτο τμήμα. Α, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 82 τμήμα. Άρχεται. Τέλος. Συμβαστική 7, πρώτο τμήμα. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπο, ε, συμβαστική 7, δεύτερο τμήμα. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 84, πρώτο τμήμα. My apologies, colleagues. Συνάδελφε, ζητώ συγγνώμη. Δεν είναι τροπολογία 84, είναι η συμβιβαστική 8. Συμβιβαστική 8 ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Amendment 84, the first part. The vote is τροπολογία 84 πρώτο τμήμα άρχεται. The vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 84 δεύτερο τμήμα που είναι ονομαστική κλίση άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 87. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 89. Άρχεται. Closed. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 90. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 91. Άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 92. Πρώτο τμήμα. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 92, δεύτερο τμήμα, άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 93. Όχι, συγγνώμη, συνάδελφοι. Συμβαστική 9, άρχεται. Συμβαστική 9, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 94 άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται τροπολογία 95, άρχεται. Τέλος εγκρίνεται. Τροπολογία 97 άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 98 άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 99 άρχεται. Τέλος εγκρίνεται. Τροπολογία 100. Τέλος. Εγκρίνεται. 101. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. 102. Άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. 103. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. 104. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 105. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 107 άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 108 άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. 110 άρχεται. Τέλος. Έγκρινεται. Συμβαστική 10 άρχεται. Τέλος. Έγκρινεται. Τροπολογία 112 άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. 113 άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. 115 άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. 100... 16. 15 είπε ο Πρόεδρος, αλλά την κάναμε 116. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Τώρα είμαστε στα συλλογικέ σκέψεις. Τροπολογία 1. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Μπορούμε να τις κάνουμε μπλοκ. Τι λέτε. Μέχρι και την 7. Unblock. Ναι, σύμφωνοι. Τροπολογίες λοιπόν 3 μέχρι και 7 άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Ε, άρχεται. Τέλος, εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Τέλος, εγκρίνεται. 14. Άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. 15. Ε, Τέλος. Απορρίπτεται. 17. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. 18. Τέλος. Απορρίπτεται. 19. Τέλος. Απορρίπτεται. 20. Ε, Άρχεται. Τέλος. Τροπολογία 21. Άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. 22. Άρχεται. Τέλος. Έγκρινεται 23, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2, πρώτο τμήμα, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2, ε, δεύτερο τμήμα. Τέλος. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας ε, ε η τροπολογία 32 άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 31 ψήφοι υπέρ. Προς 18 κατά. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε αμέσως στο επόμενο θέμα. Επόμενη ψηφοφορία. Έκθεση για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Άρθρο 116, παράγραφος 7 του κανονισμού για την περίοδο 2014 έως 2015. Η συγγήτρια είναι η κυρία Λάουρα Φεράρα. Λάουρα, θα ήθελα το λόγο ή να περάσουμε αμέσως στη ψηφοφορία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές για την πολύτιμη συνεισφορά τους ε, σε αυτή την έκθεση. Ε, εύχομαι σήμερα να εγκριθεί αυτή η έκθεση, γιατί ε, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εγγυηθεί τη διαφάνεια, τη συμμετοχή των πολιτών, θέλει να εγγυηθεί την απολοποίηση στην πρόσβαση των εγγράφων των ευρωπαϊκών θεσμών Θέλει δηλαδή να εξασφαλίσει τη συμμετοχή σε όλες τις φάσεις της νομοθετικής διαδικασίας και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Γι' αυτό ευχαριστώ και πάλι τους συνεισηγητές και καλή ψήφο. Σα ευχαριστώ πολύ. Α περάσουμε αμέσω στην ψηφοφορία. Συμβαστική πρόταση 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Άρχεται. Το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίσατε όλοι. Υπάρχει κάποια καθυστέρηση με το ηλεκτρονικό σύστημα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 22. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Πρώτο τμήμα. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Πρώτο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 43. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 7 μπις άρχεται, πέρας, εγκρίνεται. 49 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. Τροπολογία 52 άρχεται. Πέρας, Απορρίπτεται. Τροπολογία 53. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 56. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 55. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 8. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 9. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 63. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 62. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 65. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 71. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 73. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 9 πις. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 78. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 79. Άρχεται. Συνάδελφοι, δεν έπρεπε να έχουμε ψηφίσει την 79. Ακυρώνεται αυτό γιατί καταπίπτει πλησία. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 80. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 81. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 83. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτωται. 82. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 90. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 91. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 92. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 93. Άρχεται. 93. Πέρας. Εγκρίνεται. 94. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 95. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 96. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 97. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 98. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Υπομονή, το επόμενο θα είναι δύσκολο. 99, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 100, άρχεται. Πρώτο τμήμα. Πέρας. εγκρίνεται. 100 δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 101 πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 102. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 103. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 104. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 106. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 107. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 108. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 109. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 110. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 111. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 112. Ε, Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 113. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 και 8 είναι ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε unblock την 3 έως 7. Ωραία. Τροπολογίες 3 έως 7 στις θεολογικές σκέψεις. Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Με συγχωρείτε. Ήμουν αισιόδοξο περιβολικά. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. 1. Τροπολογία 1. Γιούρι. Λοιπόν, συνάδελφοι, ψηφίζουμε τις ε, τέσσερις παραγράφους. Πρώτη παράγραφος, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3, Γιούρι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ονομαστική, άρχεται. Εγκρίνεται με 45 ψήφους υπέρ, μία κατά συγχαρητήρια στην συγγήτρια. Last vote before you go. Colleagues, let's just get down to it. It's on the follow-up to the Parliament. σε ό,τι αφορά το ψήφισμα της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 11 Φεβρουαρίου 2015 σε ό,τι αφορά τη χρήση βασανιστήριων από τη CIA. Εγώ είμαι ο εισηγητής και δεν θέλω να πω τίποτα πριν από την ε, ψηφοφορία. Τροπολογία 33. Έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 34. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 35. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Έγκρινεται. 36. Έναρξη. Πέρας. εγκρίνεται. 37 έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 38 έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Συγγνώμη, ε, έναρξη ψηφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 40. Ε, έναξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 41. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 42. Ψηφίζουμε. πέρασε. Εγκρίνεται. 43. Πρώτο τμήμα. εναρξε Πέρας. Απορρίπτεται. Σαράντα έξι. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 47 και 48 και 49. Από κοινού. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται 50. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 51. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 52. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 53. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 57, 58 και 59. Ταυτόσημες. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 60. Ψηφίζουμε. Πέρας εγκρίνεται 61, 62 και 63 ταυτόσημες έναρξη. Εγκρίνεται. Μάλλον, ναι, πέρασε και εγκρίνεται. 64 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 65. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 66. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 67, 68, 69 ταυτόσημες. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 70. Πέρας. Εγκρίνεται. 71. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 72. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 74 ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε την 74 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 75 πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Συγγνώμη, μόνο το δεύτερο τμήμα, συνάδελφοι. τη 75 θα ψηφίσουμε. 75, δεύτερο τμήμα, παρακαλώ, ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 76. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 77. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 78. Ψηφίζουμε. Η 81. Πρώτο τμήμα. Έναρξη παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 81. Δεύτερο τμήμα τώρα ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 82. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 83. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 84. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 85. Έναρξε. Πέρας. Εγκρίνεται. 86. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 4 και 5 είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ψηφίζουμε. Αν ε, συμφωνείτε, εγκρίθηκε η έξε. 7 έως 11. Αν δεν έχετε αντίρρηση μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί. Ναι, κουράζεστε. 7 έως 11 unblock. ψηφισμα περας Πέρας. Εγκρίνονται. 12-13. Ταυτόσημες. Ψηφίσμα. Πέρας. Και αυτές εγκρίνονται. Οι 14 ψηφίζουμε. Πέρας. 15 ψηφίζουμε. Συγγνώμη, εγκρίθηκε. Οι 15 τώρα λοιπόν ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 16 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 17. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 21. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 22. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 23. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 24, 25 και 26. Α, συγγνώμη, 24. Ψηφίζουμε την 24. Έχει σπορθεί. Καταλαβαίνετε. Πέρας. Απορρίπτεται. 25 και 26 είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 29. Ή 29. Ή 27. 27. Συγγνώμη, ή 27. Ψηφίσουμε παρακαλώ τον 27. Πέρας για τον 27. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 29, 28. 29, 29 ψηφίσουμε παρακαλώ την 29. Πέρασε. Απορρίπτεται 30. Ψηφίζουμε και τώρα πέρασε. Εγκρίνεται 31. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο παρακαλώ στο σύνολό του έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Κύριε Ζολή, θέλετε να πάρετε το λόγο, είναι μια διευκρίνηση. Θα ήθελα να μας επαναλάβετε κατά πόσο η τροπολόγη 77 εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε. Η 77, ρωτάει ο πρόεδρος, διαγραφή της παραγράφου 13 Εγκρίθηκε, εγκρίθηκε, λέει ο πρόεδρο. Εντάξει. Δεν ξέρω κατά πόσον πήγα πολύ γρήγορα. Τροπολογία 13, 77, παράγραφος 13, η διαγραφή εγκρίθηκε. Ήταν σαφές. Δεν διευκρίνησα ότι πρόκειται για διαγραφή. Είπα ότι ήταν απλά η τροπολογία 77. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κατανοητό από όλους. Αν ε, α, αυτό θα καθορίσει την τελική σας ψηφοφορία, να το διευκρινίσουμε ασφαλώς. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ας ψηφίσουμε λοιπόν το τροποποιημένο κείμενο έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, παρακαλώ. Πέρας. Τώρα πέρας. Εγκρίνεται 27 η ψήφη υπέρ μία αποχή. Σας ευχαριστώ πολύ και έτσι ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες μας. Colleagues, are moving immediately to the next points on the agenda. Και πάρα αυτά περνάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ να κάνετε ησυχία. Εξερχόμενοι τις εκούσες. And we are moving immediately. Και έτσι περνάμε κατευθείαν στο σημείο 11 colleagues, we, we're short. Συνάδελφοι, δεν έχουμε χρόνο. Αν θέλετε να φύγετε, παρακαλώ να κάνετε ησυχία, γιατί θέλω να συνεχίσω με δύο σημαντικά ζητήματα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Στο 11 έχουμε φτάσει για τα προσωρινά μέτρα στον τομέα διεθνού προστασία υπέρ τη Σουηδία, σύμφωνα με το άρθρο 9 τη απόφαση του Συμβουλίου 2015-2023 και σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης του Συμβουλίου 2015-1601, Σκακέλερ, η συγκεκριά. Πρόκειται για έξεταση του σχεδίου έκθεσης και θα ορίσουμε και την Προθεσμίας κατάθεσης τροπολογίων 15 Δεκεμβρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση για την προσωρινή αναστολή της Σουηδίας από το μηχανισμό αν επανεκατάσταση όπω ε, αποφασίστηκε από τι αποφάσει του Συμβουλίου 2015-2023 και 2015-2016-01. Σύμφωνα με το άρθρο 9 των αποφάσεων αυτών, ένα κάθος μέλος μπορεί να ανασταλεί από τη συμμετοχή στο μηχανισμό αυτό, όπου είναι αυτό ενδεδειγμένο, αν υπάρχει ξαφνική εισρωή υπηκών τρίτων χωρών. Κυρία Σκακέλερ, είστε η συγγήτρια και θα μας παρουσιάσετε το σχέδιο της έκθεσης και τώρα θα της δώσω το λόγο και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τους συναδέλφους. Κυρία Σκακέλερ, παρουσιάστε παρακαλώ εν συντομία το σχέδιο έκθεσης. Και πριν ξεκινήσετε, συνάδελφοι σας παρακαλώ ησυχία. Thank you very much. And first let me also thank uh, the shadow rapporteurs for the very kind and constructive cooperation. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ τους και για την επικοδομητική του συνεργασία σε αυτό το θέμα. Όπως ήδη αναφέραμε, κάνουμε αυτή την έκθεση γιατί η Σουηδία έστειλε δύο επιστολές ε, στην Επιτροπή στις 5 Νοεμβρίου ε, ε, ζητώντας να γίνει δικαιούχος ε, του προγράμματος με την μετεγκατάστασης. Ε, είπαμε λοιπόν το ένα έτοιμο ήταν να είναι δικαιούχος και το άλλο να εξαιρεθεί. Και μιλάμε για την, ε, με την μετεγκατάσταση, το σχέδιο εκείνο που ορίστηκε πέρυσι. Θυμάστε ότι είχαμε δουλεύσεις εδώ. και μιλήσαμε, είχαμε την πρόταση της Κομισιόν 15 Δεκεμβρίου 2015 που μιλάει για 120.000. Δεν είναι εξαίρεση λοιπόν για τους 160.000, από τους 160.000 γιατί οι 160.000 με κατάσταση είναι δύο κομμάτια, 40.000 και 80.000. Και δεν μιλάμε για τις 120.000. Για να καταλάβετε σε προσωρινή ε, εξαίρεση από την ε, μετεγκατάσταση ζητήθηκε λοιπόν και η Αυστρία. Αλλά το Κοινοβούλιο διαβουλεύεται και δίνει γνωμοδοτή μόνο για τη Σουηδία και όχι για την Αυστρία. Ε, δεν ξέρω γιατί και μην με ρωτήσετε. τώρα δεν υπάρχει άλλο αίτημα. Η προθεσμία για την υποβολή τέτοιου αιτήματος ήταν 26 Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου. Τα κράτη-μέλη μπορούν μέχρι φέτος το Σεπτέμβριο να, γίνουν να ζητήσουν να γίνουν δικαιούχοι για την, μετεγκατάσταση. Ναι, την κατάσταση. Αυτά λοιπόν ως ιστορικό. Θα πρέπει να πω επίσης ότι υπάρχει πρόταση της Κομισιόν για το πώς θα αντιμετωπιστεί το σουηδικό αίτημα και η Κομισιόν προτείνει να εξαιρεθεί η Σουηδία από την κατάσταση για ένα χρόνο αλλά να μην γίνει ε, δικαιούχος της ε, μετεγκατάστασης. Αυτή είναι η πρόταση της Κομισιόν, τη στέλνει στο Συμβούλιο. Ξέρουμε ήδη πως το Συμβούλιο έχει μεγάλη πλειοψηφία υπέρ ε, της πρότασης της Κομισιόν και ότι το κάνουνε. Ωστόσο πρέπει πάλι να γνωμοδοτήσουμε. Τύπηση. Αυτό μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, είτε να το εγκρίνουμε την πρόταση της Κομισιόν, είτε να την απορρίψουμε βασικά. Αυτές τις επιλογές έχουμε. Και η Σουηδία, όπως γνωρίζουμε, απετέλεσε πάντα πρότυπο γιατί εφάρμοσε καλύτερα το νόμο περί ασύλου, έχει δεχτεί περισσότερους πρόσφυγες από τα άλλα κρατημέλη, ήδη όταν πολλοί Σύριοι έφταναν. Η Σουηδία έδωσε άμεσα άδεια ώστε να μείνουν οι Σύριοι με πολύ καλές συνθήκες υποδοχής, ε, οι προδιαγραφές και για τους μη συνοδευόμενους ανήλικους ε, ήταν εξαιρετικές. Και ε, πιστεύω πως τα άλλα θα έπρεπε να παραδειγματιστούν από τις συνθήκες εκεί. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια παράπονα από άλλα κρατημέλη, των οποίων ε, τα συστήματα ασύλου πιέζονται και αυτό ισχύει ό,τι σύστημα ασύλου και αν Ακόμα και στην Σουηδία που ήταν καλά το σύστημα ασύλου, πάλι πιέζεται γιατί τόσοι πολλοί πρόσφυγες πήγαν εκεί. 163.000 πρόσφυγες νομίζω έφτασαν μόνο πέρυσι στη Σουηδία. Και εμείς ως η ομάδα των σκιωδών ε, είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων στις 16 Μαρτίου, ακριβώς πριν από την προθεσμία κατάθεσης ε, της έκθεσης. Θέλαμε να ακούσουμε και την άποψη των Σουηδών εμπειρογνωμόνων και κάναμε μια τέτοια συνάντηση με εκπροσώπους των Σουηδικών τοπικών αρχών και των, ε, ε της υπηρεσίας ασύλου και μετανάστευσης. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ενημέρωση για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η ε, Σουηδία. Προσωπική μου σύσταση θα ήταν και αυτό προτείνω και στην έκθεση να μην ακολουθήσουμε την πρόταση της Κομισιόν για εξαίρεση της ε, Σουηδίας για ένα χρόνο λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια προσπάθεια που έχει καταβάλει η Σουηδία και λαμβάνοντας υπόψη και τις προκλήσεις που έχει ε, με τον τεράστιο αυτό αριθμό ε, προσφύγων. Ωστόσο δεν είναι σημαντικό να ζητήσουμε από την Σουηδία να επεγκαταστήσει τον κόσμο που πρέπει από αυτές τις 120.000. Είναι αλήθεια ότι η Σουηδία έχει μείνει μόνη της, ενώ τα άλλα κρατημέλη δεν έχουν κάνει το δικό τους μερίδιο δουλειάς, δεν έδειξαν αλληλεγγύη όπως η Σουηδία. Γι' αυτό και πιστεύω ότι τώρα που υπάρχει ο μηχανισμός αλληλεγγύης, θα ήταν παράξενο να πούμε τώρα ότι ε, τώρα μπορεί η Σουηδία να φύγει από το μηχανισμό αλληλεγγύης. Ενώ θα έπρεπε να χρησιμεύσει ως πρότυπο για να ακολουθήσουν και άλλα μέλη το δρόμο αυτό. Τώρα έχουμε 130.000 πρόσφυγες. Στη Σουηδία, η Σουηδία ζήτησε να μετεγκαταστήσει 567 από την Ιταλία και 1830 από την Ελλάδα. Ε, από την Ιταλία 567 και από την Ελλάδα 1830. Για, σε δύο χρόνια, αν και η Σουηδία υπόκειται σε μεγάλη πίεση. Πιστεύω πως αυτά τα νούμερα δεν είναι και πολύ υψηλά, ότι μπορούν να τα χειριστούν στην, στην Σουηδία, δηλαδή, γιατί έχουν εξαιρετικές υπηρεσίες και εξαιρετικούς ανθρώπους που συναντήσαμε και πολλούς ακόμα που εγώ προσωπικά συνάντησα, αλλά που εσείς βεβαίως του γνωρίζετε καλύτερα. Αυτή, τα νούμερα δεν είναι και τεράστια. Είναι πολύ συμβολικό κατά νούμερα και να πούμε λοιπόν ότι αυτοί οι μηχανισμοί αλληλεγγύης θα πρέπει να ισχύσουν για όλους και δεν πρέπει να αρχίσουμε με τις εξαιρέσεις. Έχαμε βέβαια τη δυνατότητα να πούμε τη γνώμη μας για την αυστριακή υπόθεση, αλλά, για την σουηδική περίπτωση, αλλά όχι για την αυστριακή. Ε, δεν κατάλαβα κανείς γιατί. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι έχουν τα πράγματα. και στην αρχική έκθεση έτσι είπαμε ότι τα νούμερα είναι μικρά, ότι αυτή θα είναι μόνο η αρχή και τώρα θα είναι σωστό να πούμε ότι όλοι πρέπει να τηρήσουμε το σύστημα και να μην αρχίσουμε τις ε, παρακλήσεις και τις παρακάμψεις. Εξάλλου η Κομισιόν έχει ανακοινώσει νέο προσαλλαγές για το σχέδιο με την κατάσταση. Θέλουν τις θέσεις της Ουγγαρίας που υποτίθεται θα ήταν δικαιούχος ε, αλλά είπε ότι δεν θέλει να είναι δικαιούχος αυτές οι θέσεις τώρα θα προτείνει η Κομισιόν να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις θέσεις και να μετατρέψουμε σε ένα σχέδιο αϊκούσιας με την κατάσταση, αλλά και να επιτρέπουν στους φοιτητές να σπουδάζουν στην Ένωση να δίνουν και άδειε εργασία από τους 50.000 ανθρώπους. 50.000 άνθρωποι. Ε, θα γίνει ένα νέο πάλι πρόγραμμα. Έχουμε ξεκινήσει επίγουσε δικασίες, έχουμε δεχτεί ότι δεν μας διαβουλεύθηκαν, ότι στο μέλλον θέλουμε να έχουμε σωστή διαβούλευση και ότι, όπως είπα, δεν θα πρέπει να ρίξουμε νερό στο κρασί μας. Τα νούμερα είναι μικρά. Ε, και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη θα τηρήσουν τη συμφωνία. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ τους Κιώδης και ελπίζω πως θα μπορέσουμε να συζητήσουμε θετικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρος, ευχαριστώ. Σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Έχουμε επίσης να συζητήσουμε και το θέμα του κυρίου Κέρκοπ για το έκρης μέχρι τις 12.30. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Είναι λεπτό το ζήτημα εδώ, ευαίσθητο και πρέπει να ακούσουμε την άποψη όλων των σκιωδών εισηγητών. Η θέση της εισηγήτριας ήταν ξεκάθαρη. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω όλους εσάς, αλλά σας παρακαλώ να συνοψίσετε και να είστε όσο το δυνατόν σαφέστεροι. Αρχίζουμε με την σκιώδη του ΕΛΚ, κυρία Αναμαρία Κορατζαμπίλτ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως είπε και η Κέλλερ, η Σουηδία έχει μείνει μόνη της εδώ. Το, τα συμπεράσματα όμως που έβγαλε είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να, να δεχτώ. Είναι απαράδεκτα και δικαιολόγητα. Τα επιχειρήματά της είναι ε, για μένα κάτι που δεν μπορώ να δεχτώ, διότι η Σουηδία θα έπρεπε να λάβει υποστήριξη. Ήταν δυσανάλογη η αλληλεγγύη που έδειξε η ίδια η Σουηδία και δυσανάλογος ο ε, φόρτος που έπρεπε να επομιστεί. Έχουμε πολλά μέσα στη διάθεσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξουμε τις χώρες που δέχονται μεγάλη πίεση, τη Frontex ε, και άλλες. Και τα νούμερα έχουν ως εξής. 7.330 ένα παιδιά, πολλοί ασυνόδευτοι ανήλικοι. Στην Σουηδία βρίσκονται οι περισσότεροι ασυνόδευτοι ανήλικοι από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί αρχίζω τώρα με τα παιδιά και τους ασυνόδευτους ανήλικους. Γιατί τα κράτη-μέλη πρέπει να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν το γεγονός ότι η Σουηδία φέρεται ε, έτσι όπως ε, πρέπει να φέρονται όλοι. Και μην ξεχνάτε ότι οι ανήλικοι χρειάζονται πολύ περισσότερους πόρους έτσι ώστε να τους παρέχονται αυτά που πρέπει. Η Σουηδία επίσης έχει 143.000 εκρεμεί αιτήσει ασύλου. Ο προϋπολογισμός ε, για τη στέγαση είναι 600 δισεκατομμύρια σουηδικέ κορώνες. Είναι μεγαλύτερος από τον ε, αμυντικό προϋπολογισμό της χώρας. Διπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός ε, της υπηρεσίας μετανάστευση. Και μας έχουν ενημερώσει 60 δήμοι ότι δεν αντέχουν άλλο. 163.000 το 2015, αντίστοιχη το 2016. Το Νοέμβριο η Σουηδία ε, δεχόταν 11.000 ανθρώπους την εβδομάδα. Και η Σουηδία είναι μια χώρα πρώτης υποδοχής, διότι πολλοί ε, που έρχονται στην Σουηδία δεν έχουν καταγραφεί πουθενά αλλού. Η Σουηδία λοιπόν πρέπει να διαθέσει τους πόρους για την τελική ένταξη στο σχολείο, στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο ε, σύστημα ε, ιατρικής περίθαλψης, αλλά και πόρους ε, για να καταγράψει δακτυλικά αποτυπώματα, για να κάνει όλες αυτές τις εργασίες που χρειάζονται για τις περιπτώσεις πρώτης εισόδου. Και δεν βλέπω κανένα άλλο τρόπο να στηρίξουμε ένα κράτος που δέχεται τόσο πολύ πίεση ό,τι και να κάνουμε, όσο περισσότερους πόρους και να διαθέτουμε για τους ε, πρόσφυγες, ε, δεν μας ακολουθεί κανείς, δεν το εκτιμά κανείς αυτό και η ε, Αυστρία, εδώ μόλις ακούσαμε, πώς, δεν συμπερι... πώς αρνείται να συμμορφωθεί, να δείξει αλληλεγγύη. Ήμασταν οι πρώτοι που δεχθήκαμε πρόσφυγες από την Ερυθρέα. Είμαστε η χώρα που διαθέτει περισσότερα χρήματα από όλου στο Ταμείο για τους Πρόσφυγες, στο Ταμείο για τη Συρία. 64% του Ταμείου για τους πρόσφυγες ε, χρηματοδοτείται από τη χώρα μου, από τη Σουηδία. Και αυτό που λαμβάνουμε ως απάντηση είναι ποιο. Ότι θα σας τιμωρήσουμε ακριβώς επειδή είσαστε τόσο καλοί στη δουλειά σας. Όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή ε, θα έχουν καλύτερη μεταχείριση από εσάς. Επειδή εσείς είστε τόσο καλοί δεν χρειάζεται καμία βοήθεια. Έτσι λειτουργεί η αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή μήπω οι χώρες οι οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να αναπτύξουν ε, μεγαλύτερη χωρητικότητα, για να καταρτήσουν ανθρώπους, για να δημιουργήσουν ένα λειτουργικό δίκτυο ε, για την μετανάστευση να εφαρμόσουν τους νόμους που δεν τους εφαρμόζουν, αυτές έχουν τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι φυσιολογικό, κυρία Κέλλερ. Εγώ το θεωρώ απαράδεκτο, εξοργιστικό και το θεωρώ ταπεινωτικό για τον Σουηδικό λαό, ο οποίος ήταν εκεί κάθε μέρα, ερχόταν στους δρομικού σταθμούς, έδινε νερό, ήταν εθελοντές, βοηθούσαν με όποιο τρόπο μπορούσαν. Και ποιος είναι ε, ο τρόπος αντιμετώπισης, του στέλνετε στο διάβολο. Η κυρία Σκακέλερ θα έπρεπε να μην ξεχνά πως είναι μέλος των Πρασίνων και η κυβέρνηση της Σουηδίας είναι συνασπισμός Πρασίνων και Σοσιαλιστών. Αυτό που ζητήσαμε είναι αναστολή για ένα χρόνο, όχι να μην δεχτούμε κανέναν άλλον πρόσφυγα, όχι να κλείσουμε τα σύνορα. Έχουμε περίπου 700 πρόσφυγες που φτάνουν στη Σουηδία κάθε μέρα. Αυτό που ζητούμε είναι μια αναστολή για ένα χρόνο έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε πρόσφυγες και να διατηρούμε το υψηλό επίπεδο βοήθεια που παρέχουμε μέχρι τώρα. Αυτό που ζητούμε είναι να μας βοηθήσετε να μην ρίξουμε αυτό το επίπεδο, να μας δώσετε λίγο χρόνο έτσι ώστε να ε, επανέλθουμε από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης ε, στην οποία λειτουργούν οι υπηρεσίες μας σε μια αξιοπρεπή κατάσταση. Αυτό που γίνεται τώρα είναι απαράδεκτο, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ζητήσω να απορρίψετε και να καταψηφίσετε την έκθεση Κέλλερ. Okay, um, Um, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στους σοσιαλδημοκράτες και θα δώσω το λόγο στην κυρία Αναχέντη, η οποία θα μιλήσει εκ μέρους της ε, σκιώδη δούσης Όχι, κυρία Ζίπελ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα αρκετά συναισθηματικό. Εγώ θα ήθελα να δω μια πιο ψυχρή και αντικειμενική συζήτηση, γιατί όπως είπε και ο Πρόεδρος είναι πολύ λεπτό και βάστη το ζήτημα. Και μέχρι ένα σημείο συμφωνώ με το σκεπτικό της κυρίας Κέλλερ και αναφέρομαι δηλαδή στο ότι η κατάσταση στη Σουηδία έτσι όπως έχει σήμερα έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με την κατάσταση στην Ελλάδα. Και ας μην ξεχνάμε ότι η παρούσα κυβέρνηση της Ελλάδας δεν ευθύνεται για όλα όσα δεν έχουν γίνει ή έχουν γίνει τα περασμένα χρόνια στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν καταλαβαίνω απόλυτα μέχρι ενός σημείου ότι αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιστροπής δεν μπορεί να στηριχθεί. Από την άλλη όμως, Συμφωνώ και με το ότι τα τελευταία χρόνια η Σουηδία σε σχέση με τον πληθυσμό της έχει υποδεχτεί τους περισσότερους ε, πρόσφυγες από όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και είναι ακόμα πρόθυμοι να συνεχίσουν να δέχονται πρόσφυγες. Το μόνο που ζητούν δηλαδή είναι ένας χρόνος ε, προθεσμία έτσι ώστε να μπορέσουν να ε, ξαναχτίσουν τις υποδομές τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν να υποδέχονται μετανάστες. Γι' αυτό λοιπόν ε, συμφωνώ με την στήριξη της ιδέας της Επιτροπής. Δεν θέλω όμως να ρίξω το βάρος στην Ελλάδα. Θέλω να ρωτήσω γιατί ορισμένα κρατημέλη είναι απόντα, δεν δείχνουν καμία απολύτως αλληλεγγύη, δεν έχουν καμία απολύτως ε, πρόθεση να δεχτούν πρόσφυγες, να στείλουν προσωπικό για στήριξη στην Ελλάδα, να διαθέσουν χρήματα για επικούς τρίτο, ε, τρίτων χωρών, να στείλουν βοήθεια σε τρίτες χώρες για να στηρίξουν την προσπάθειά μας. γιατί δηλαδή κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέχουν παντελώς από αυτό που συμβαίνει τώρα με το μεταναστευτικό ζήτημα και με τους πρόσφυγες που ζητούν άσυλο. Τέλος τι μήνυμα θέλουμε να δώσουμε, τι μήνυμα δίνουμε με τη μία ή την άλλη απόφαση. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που θα κάνουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε που θα στηρίξει τις προσπάθειές μας και να δείξουμε ευαισθησία. Πρέπει να εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή όλα τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών και να μην ξεχνάμε επίσης ότι πρέπει να εργαστούμε έτσι ώστε στο μέλλον να βελτιώσουμε τις συνθήκες στην Ευρώπη, έτσι ώστε όχι μόνο η Σουηδία να είναι η χώρα που θα δέχεται τους περισσότερους ετούντες άσυλο, όχι μόνο η Μάλτα ή η Γερμανία, αλλά να συμφωνήσουν όλα τα κρατημέλη να δεχτούν ετούντες άσυλο, να δεχτούν πρόσφυγες, να τους φροντίσουν και όχι να χτίζουν φράχτες και να κλείνουν σύνορα για να κρατήσουν τους ανθρώπους αυτούς εκτός. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό, όχι μόνο για τη Σουηδία, αλλά και για τους υπόλοιπους. Ο κύριος ε, Κέρκο θα μας δώσει την άποψη της ε, ομάδας ECR τώρα, γιατί θα λείπει το απόγευμα. Ε, μετά η κυρία Μπιόρκ, σκιώδη ηγήτρια, η κυρία Βίνμπεργκ και ο κύριος ε, Τζαντόφσκι και η κυρία Χολμάιερ θα λάβουν το λόγο. Ξέρω πως ε, δεν είμαι ίσως δίκαιος, αλλά σας παρακαλώ να είστε πολύ πολύ σύντομοι. Δεν θα μείνει χρόνος για τον κύριο Κέρκοπ αλλιώς. Παρακαλώ περιοριστείτε στα ένα ή δύο λεπτά. Και μείνετε εντός θέματος. Προσωρινός μηχανισμός μεταγκατάστασης και ο ρόλος της Σουηδίας στην προσφυγική κρίση. Αυτό συζητάμε τώρα. Η κυρία Μαλίν Μπιόρκ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από πλευρά της GoNGL υποστηρίζουμε τον εισηγητή και ως ε, Σουηδή ξέρω ότι έχουν γίνει προσπάθειες Έχω δει την αλληλεγγύη. Έχουμε άτομα εδώ στην αίθουσα που ήταν ε, στους διδρομικούς σταθμούς και δεν τους ε, γελιοποιεί το γεγονός ότι δεν θα συμπεριληφθεί η Σουηδία στο μηχανισμό. Αυτό που τους γελιοποιεί είναι ότι δεν ανταποκρίνονται στην αλληλεγγύη τους όλα τα πολιτικά κόμματα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τους γελιοποιεί, όχι η κατάσταση αυτή. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο το ότι χρησιμοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι που είναι στους σταθμούς δρομικού ως επιχείρημα. Η Σουηδία έχει να λάβει μεγάλο τμήμα της ευθύνη αφετέρου. Και αυτό νομίζω το γνωρίζουν όλοι εδώ στην αίθουσα. Αν το σουηδικό σύστημα πρόνοιας δεν ε, θα πέσει. Πολύ αλληλεγγύη είδαμε και πολύ επαγγελματισμό και με τον τρόπο αυτό θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στη Σουηδία η πρόνοια και οι δυνατότητε απορρόφησης της Σουηδία υποστηρίζονται με 35 εκατομμύρια από το ΑΜΥΦ. Αν έχουμε τέτοια ελλείμματα στη Σουηδία, στο κράτος πρόνοιας, είναι δικό μας ε, ζήτημα. Είχαμε περικοπές στη φορολόγηση των πλουσίων, είχαμε προβλήματα στην ε, ε, φορο... στην σε ό,τι αφορά το φορολογικό μας σύστημα, τα δικά μας ελλείμματα είναι αυτά που φτάνουν. Δεν μπορώ να δεχτώ οποιοδήποτε επιχείρημα που λέει ότι η υποδοχή προσφύγων αποτελεί τιμωρία. Δεν έχω κάνουν τίποτα να συζητήσω με τέτοια άτομα που χρησιμοποιούν τέτοια επιχειρήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση και είναι και πάρα πολύ ευαίσθητη, γιατί αυτό θα διαμορφώσει τη Σουηδία στο μέλλον και την Ευρώπη στο μέλλον. Η Σουηδική κυβέρνηση προσπαθεί να ασκήσει πίεση στις άλλε χώρε για να αναλάβουν τι ευθύνε. του. Το αναγνωρίζω αυτό, πιστεύω ότι είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι σωστό αυτό ο τρόπο. Το Δουβλίνο θα πρέπει να τροποποιηθεί, η μετεγκατάσταση θα πρέπει να λειτουργήσει και για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να καταδείξει η Σουηδία ότι συμμετέχει 100% και ότι ε, δεν θα αυτοεξαιρεθεί. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος, και πολύ λυπάμαι που σας ε, ζητώ να είστε σύντομοι. Σας παρακαλώ, το ένα λεπτό προσπαθείτε να τηρήσετε ως ε, χρόνο ομιλίας, γιατί έχουμε και ένα θέμα για την τρομοκρατία στη συνέχεια. Ο κύριος, ε, ο εκπρόσωπος του ECR, παρακαλώ, προσπαθείτε να τηρήσετε το όρο των ε, ενός-δύο λεπτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος, μιας και το ζητάτε, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε μία απόφαση ευνοϊκή προς το αίτημα της Σουηδικής κυβέρνησης, μια και το ζητάει η Σουηδία, ζητά προσωρινή αναστολή. Δεν ε, μιλάει για υπονόμευση του συστήματος επανεγκατάστασης, όχι. Προσωρινή αναστολή ζητάει. Θεωρώ ότι υπάρχουν λόγοι που οθούν τη Σουηδία στην υποβολή τέτοιου αιτήματο και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε όλες τις προσπάθειες που καταβάλει η Σουηδία για να υποδεχτεί τους ε, μετανάστες. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την ε, άριστη συμπεριφορά της στον τομέα αυτό και θα πρέπει να θεωρώ να δείξουμε εμπιστοσύνη στο Συμβούλιο και στην απόφαση της θεωρώ ότι θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μην είμαστε δογματικοί στην τοποθέτησή μα. Α μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η ουσιαστική κυβέρνηση πάντα καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την υποδοχή των μεταναστών. Αυτά για την κυρία Κέλλερ για να επιδείξει μεγαλύτερο πνεύμα ευελεξίας. Ο πρόεδρος, η φιλελεύθερη, κύριε Ντεπρέ, ένα λεπτό αν θέλετε για να μας παρουσιάσετε και τις δικές σας θέσεις. Σύντομα, Πρόεδρε. Δεν είμαι σκιώδης για το θέμα αυτό, αλλά παρόλα αυτά θα πάρω το λόγο εξ ονόματος της ομάδας μου. Για να εκφράσω ξα... καταρχής το πώς εκτιμάμε τους ειδούς και τα όσα έχουν κάνει για τους μετανάστες. Έχει κάνει, έχουν κάποια πολλά από αυτά που τους αναλογούσαν. Και αν ε, ζητούν ε, μια τέτοια πάυση, μια προσωρινή αναστολή, δεν βλέπουμε ποιο ηθικό με υπόβαθρο μπορούμε να τους πούμε ότι δεν το δικαιούνται. Δεν θα ήθελα λοιπόν να ακολουθήσουμε την εισηγήτρια στην επιχειρηματολογία της και προσωπικά εδώ θα ήθελα να επιδείξουμε πνεύμα ανθρωπισμού και κυρίως να μην ε, δίνουμε μαθήματα σε όσους έχουν κάνει τη δουλειά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη θέση σας και για την συντομία σας, κυρία Ντεπρέ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Άννα Χέντ. Και πάλι σας ζητώ συγγνώμη που σας πιέζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι η εξαίρεση για τη Σουηδία είναι σημαντική για δύο λόγους. Αν στο Κοινοβούλιο θέλουμε να έχουμε ένα κοινό σύστημα ασύλου, με ένα δίκαιο σύστημα ανακατανομής η χώρα η οποία έχει αναλάβει τις μεγαλύτερες ευθύνες κατά κεφαλή θα μπορούσε και θα έπρεπε να πάρει μια προσωρινή αναστολή από το σύστημα αυτό. Και ο άλλος λόγος έχει να κάνει με τους συνοριακούς ελέγχους και το μέλλον του Σένιεν. Έχει μειωθεί στις τελευταίες 6 μήνες ο αριθμός των μεταναστών και των ετών άσυλο στη Σουηδία, αλλά αυτό ε, σχετίζεται με τους ε, ελέγχους στα σύνορα που έχει εισαγάγει η Σουηδική κυβέρνηση και προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι λυπηρό. Θα ήταν υποκριτικό λοιπόν από πλευρά ε, του ΕΛΚ να αντιτάσσεται στους νοριακούς ελέγχους και παράλληλα να μην κάνει και τίποτε σε ό,τι αφορά αυτό το άδικο σύστημα επανεκατάστασης. Θα υποστηρίξουμε λοιπόν μέτρα για την πιο δίκαιη κατανομή και πιο δίκαιη υποδοχή μεταναστών στην Ευρώπη. Αν ουσιαστικά αρνηθούμε την προσωρινή αυτή αναστολή, θα συνεχίσουμε τη σημερινή έλεγχη και θα αποδυναμώσουμε το Σέγγεν. Θα το καταργήσουμε. Ο Πρόεδρος, κύριε Κέρκοπ, ε, κύριε Κέρκοπ, Μπορεί να μην προλάβουμε το θέμα σας. Δεν ξέρω όμως. Θέλετε. Έχετε χρόνο άλλο, γιατί θα... ήθελετε να μιλήσετε τώρα. Α, εντάξει, όχι, να μιλήσουν και οι δύο επόμενοι ομιλητέ για ένα λεπτό. Η κυρία Βίνμπεργκ, για ένα λεπτό παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως Σουηδή, καλούμε να μιλήσω και να συνομιλήσω με μια Γερμανίδα αριστερή η οποία θα ορίσει τους νόμους για την ε, μεταναστευτική πολιτική της ε, Σουηδίας. Δεν ξέρω τι, τι να πω. Όλοι λένε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε το σουηδικό μοντέλο και πόσο καλό είναι και μετά μας μιλάτε για τους πόρους, για το προσωπικό. Ξέρετε τι συμβαίνει στη Σουηδία. Ίσως θα έπρεπε να παρακολουθείτε καλύτερα τα μέσα ενημέρωσης για να βλέπετε τι συμβαίνει. Μιλάμε για 163.000 άτομα, 163.000 άτομα τα οποία έχουν έρθει στη Σουηδία. Το τι έχει προκληθεί ε, στο σύστημα πρόνοιας, στα σχολεία, στα κέντρα υποδοχής, στη μέση του χειμώνα που ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι απελπιστική η κατάσταση. Ο κόσμος ζει στους δρόμους. Όλα αυτά τα προβλήματα. Και θα μας βγείτε εσείς να μας πείτε πόσους θα πάρουμε και αν θα, κάνουμε, αν θα πάρουμε τα προσωρινά μέτρα. Σκανδαλώδες. Η Σουηδία θα πρέπει να μπορεί να καθορίσει ποιου θα προδεχτεί και αν μπορεί να το κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό για την κυρία Χόλμαερ, λέει τώρα ο πρόεδρος. Και μετά θα ακούσουμε τον εισηγητή. Θα ήθελα να υποστηρίξω την Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ. Ε, αγαπητή Σκακέλερ, θεωρώ ότι είναι πραγματικά απαράδεκτο το γεγονός ότι μια χώρα η οποία έχει συμβάλει τόσα πολλά και ζητά αναστολή ενό έτους, ε, του, του αρνούμαστε μια στοιχειώδη βασική υποστήριξη. Αυτό ουσιαστικά ανισχύει τους ακροδεξίους ε στη Σουηδία. Θέλουμε μια λογική αντιμετώπιση των κρατών μελών. Μια χώρα η οποία έχει συμβάλει τόσο πολύ, μας απευθύνει μια τέτοια έκκληση, θα έπρεπε να ανταποκριθούμε στο αίτημά τους και όχι να το παίζουμε ηθικό διδάσκαλοι. Και θα παρακαλούσα την εισηγήτρια να αναθεωρήσει αν είναι δυνατόν την άποψή της. Ο Πρόεδρος. κυρία Σκα Κέλλερ. Αν σας δώσω το λόγο θα απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Νομίζω ότι ήταν σαφείς οι θέσεις που παρουσιάστηκαν όμως από πλευρά των διαφορών ομάδων. Ήταν λίγο πολύ σωστά οι εκπροσωπήσεις. Έχουμε την προθεσμία για την κατάθεση των προλογιών. Κάποια διαδικαστικά, αν θέλετε να θέσετε, και μετά να ολοκληρώσουμε το ζήτημα αυτό. Σας παρακαλώ. Ναι, κοιτάξτε, έχουμε διαφορετικέ απόψει ε, και αυτό είναι σωστό και εύλογο και θεμητό. Χρειαζόμαστε πιο πολύ αλληλεγγύη, σε αυτό συμφωνούμε. Απλά καταλήγουμε σε διάφορα συμπεράσματα. Ούτε θέλω να, να μου κάνετε σεμινάριο και να σας κάνω σεμινάριο για τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε εκπροσωπούμε τις κυβερνήσεις των κρατών μελών οι βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάνουν το καλύτερο για όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι ο σκοπό μα. Ασφαλώ καταλήγουμε σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτό είναι προφανέ. Επί τη διαδικασία, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να καταθέσετε τροπολογίε στην έκθεση, αλλά η καταψήφιση τη έκθεση δεν θα περάσει το σημείο σα. Κοιτάξτε, θα πρέπει να το ολοκληρώσουμε. 14 Απριλίου είναι η ημερομηνία κατάθεση τροπολογιών, η προθεσμία. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα και δεν μου αρέσει που αναγκάζομαι να σας περιορίσω, αλλά με όλο τον συναισθηματισμό των επιχειρημάτων ήταν σαφείς οι πολιτικές θέσεις της Επιτροπής. Νομίζω ότι αποτυπώθηκαν σωστά. Θα είναι σαφής λοιπόν η γραμμή των τροπολογιών. Σας είπε ποια είναι η προθεσμία. Ξέρουν και οι συγγετρία από πού θα προέλθουν, ε, από ποιο σημείο θα και έτσι λοιπόν να περάσουμε. Αναγκαστικά πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου. Έκρης. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Κερκόπ. Στις 16 Μαρτίου στη Λίμπα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μία πρόταση για να θεώρησε του έκριστου συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με υπηκόους των χωρών. Δεν θα καθυστερήσω και θα δώσω το λόγο πάρα αυτά στον κύριο Κέρκοπ για να παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης και μετά θα δούμε και τι ισχύει για την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Κύριε Κέρκοπ, έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ, συνάδελφοι, αν φεύγετε, ησύχως. Έχετε το λόγο, κύριε Κέρκοπ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σχετικά παρά τη βαβούρα μέσα στην αίθουσα, θα είμαι σύντομο, Ωστόσο, Μπορεί αυτό να είναι το τέλο τη σημερινή διάταξη για σήμερα και είναι ένα συμπληρωματικό θέμα σε κάποιο βαθμό, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό τεραστίας σημασίας, ε, διότι πιστεύω πως όλοι εδώ συμφωνούμε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών ε, εγκληματικού τύπου ανάμεσα στις δικαστικές αρχές είναι ένα βασικό στοιχείο για τη συνεργασία ε, μεταξύ ποινική ε, δικαιοσύνη ε, των 100 μελών θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη στην διασυνοριακή συνεργασία και βεβαίω στην χώρο Σέγγεν. Και γι' αυτό η έκθεσή μου στηρίζει απολύτω του στόχου τη Κομισιόν και την πρόταση που έχει υποβάλει η ίδια η Κομισιόν. Θα κάνω λίγες αλλαγές και προσθήκες εκεί όπου πιστεύω πως είναι απαραίτητες οι σωστές. Όπως είπα, στην αρχική συζήτηση που είχαμε πρόσφατα, ε, πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να επεκτείνουμε τη δυνατότητα που έχουμε για βασικούς ελέγχους για όλους όσους εργάζονται με παιδιά φυσικά και για όλους όσους εργάζονται με ευάλωτους ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων αυτών που εργάζονται στην κοινωνική πρόνοια, την υγειονομική περίθαλψη και την περίθαλψη ατόμων με ειδικέ ανάγκες καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών για ε, ποινικά δικήματα πολιτών τρίτων χωρών εκεί όπου οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν ανταλλάσσονται ανάμεσα στα κρατη ε, στην έκθεσή μου έκανα μια σαφή αναφορά ε, όσον αφορά την τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, το δικαίωμα σε δίκαια δίκη ε, και ε, κοιτάζοντας τις στατιστικές, ε, τα αιτήματα των αριθμών των αιτημάτων που γίνονται για τέτοιου είδους ελέγχους, το επίπεδο συνεργασίας και το επίπεδο ανταλλαγής των πληροφοριών ανάμεσα στα ίδια κρατημέλη, πιστεύω εντόνως, Πρόεδρε, πως μια ουσιαστική διαδικασία αναθεώρηση είναι σημαντική για τη σωστή εφαρμογή και τη σωστή νομοθεσία. Και να θυμίσω και στα μέλη πω πρόκειται βεβαίω για, για ένα εφιστάμενο επιχειρησιακό και λειτουργικό μέτρο το οποίο απλώς θέλουμε να επεκτείνουμε και σε επικόστη των χωρών. Είναι λογικό, λογική και απαραίτητη επέκταση του συστήματος. Δεν χρειάζεται δηλαδή να επανεφεύρουμε τον τροχό. Γι' αυτό και ελπίζω για γρήγορη ε, διαδικασία για να κλείσουν τα κενά, τα, τα, τα παραθυράκια που φυσικά και οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται όσο περισσότερο μπορούν. Τέλος, το έκρισε βεβαίως, όπως είπε ο Πρόεδρε, ήδη φαίνεται μάλλον παρέχει σαφώς ενδείξεις για το πώς η, διαευρωπαϊκή συνεργασία μα ε, μας βοηθά ήδη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ωφελεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες γιατί έτσι οι πολίτες μας όπου και αν βρίσκονται είναι ασφαλέστεροι. Αυτή η επέκταση βεβαίως ε, ε, ε, διευκρινίζει την κατάσταση και βεβαίως για το μέλλον απαιτεί την ενθουσιώδη συμμετοχή όλων των κρατών μελών συμπεριλαμβανομένης της χώρας μου, του Ηνωμένου Βασιλείου, σε οποιαδήποτε εξέλιξη αυτού του σχεδίου. Συστήνω λοιπόν αυτή την πρόταση και την έκθεση και προσβλέπω στις συμβολές των υπολείπων συμπεριλαμβανομένων των τροπολογιών τους, αν το θεωρούν αυτό απαραίτητο. Έχουμε μια προσωρινή προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για τις 15 Απριλίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. I think it was the 18th of April, just for the record. 18 Απριλίου είναι η προθεσμία. Ναι, ωραία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέρκοπ. Περνάμε λοιπόν τώρα στους σκιώδεις μας για αυτό το θέμα και ξεκινάμε την Anna από τους σοσιαλιστές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Καλωσορίζω τις ε, περισσότερες τροπολογίες του κυρίου Κέρκοπ πιστεύω πως θα καταφέρω να συμφωνήσω σε αυτές εγώ και η ομάδα μου. Έχω όμως μία ερώτηση που αφορά το αίτημα για πληροφορίες όταν κάποιος ε, ψάχνει δουλειά. Σε περίπτωση καταδίκης για σεξουαλικά ποινικά δικήματα δεν πρέπει να ε, εργάζεται κάποιος σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα στον τομέα της υγείας και δεν πρέπει να του επιτρέπεται να πάει σε κάποιο άλλο κράτος μέλος για να εργαστεί εκεί. Υπάρχουν 15 διαφορετικές καταδίκες και πιστεύω πως είναι ένα δύσκολο ερώτημα το ποιος δηλαδή πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Είναι κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο για το ίδιο το κράτος μέλος να κοιτάξει δηλαδή το μητρό κάποιου υπηκόου τρίτης χώρας. Φαντάζομαι ότι για τις πληροφορίες ευθύνεται το κράτος στο οποίο έχει καταδικαστεί αυτός ο επικός τρίτης χώρας. Αυτό που χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, είναι περισσότερη ε, σαφήνεια νομική σαφήνεια. Θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες. Πιστεύω επίσης πως τα δακτυλικά αποτυπώματα πρέπει να λαμβάνονται γιατί είναι αναγκαία σε ορισμένες ε, σε περιπτώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του ΕΛΚ, ο κύριος ε, Τσάρη. Örülök Σας ευχαριστούμε κύριε Κέρκοπ για την εξαιρετική σας εργασία και καλωσορίζω την ε, άποψη της ε, δεμερούς ανταλλαγής ε, πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών σε ό,τι αφορά υπηκούς τρίτων χωρών. Αυτές οι πληροφορίες θα διαβιβάζονται και σε άλλα μέλη. Θα ήθελα να ρωτήσω όμως τον Τίμωθο που κατά πόσον το σύστημα αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί και σε επικότητα χωρών που δεν έχουν ε, ε, υπηκότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι τουρίστες που έχουν διαπράξει κλίματα. Θα έλεγα λοιπόν ότι η πρόταση οδηγίας της Κομισιόν Στόχο έχει να επεκτείνει και την ε, συλλογή αποτυπω... δακτυλικών αποτυπωμάτων που είναι πολύ αποτελεσματικό μέσω εντοπίσμου. Η Κομισιόν θέλει να εφαρμόσει ένα αποκεντρωμένο σύστημα το οποίο θα ήταν πιο αποτελεσματικό από ό,τι το ισχύον αλλά κατά τη γνώμη μου ένα τέτοιο κεντρικό σύστημα θα ήταν ακόμα πιο αποτελεσματικό ακόμα και αν ήταν πιο δαπανηρό όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ πιστεύω πως δεν θα πρέπει εδώ να κάνουμε οικονομίες, γιατί ένα κεντρικό σύστημα θα μπορούσε να περιέχει όλα τα στοιχεία των 28 χωρών και θα ήταν και πιο αποτελεσματικό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα, γιατί είναι προχωρημένη η ώρα. Εγώ δεν είμαι σοσια... σκιώδης ε, των σοσιαλιστών, είναι η συνάδελφος Αναχέντα, αλλά θέλω απλά να ε, υποδείξω το ενδιαφέρον μου και τη στήριξή μου για την πρωτοβουλία της Κομισιόν και για την λογική πρόταση που θα υποβάλει ο συνάδελφος ε, Τίμωθη Κίρκοπ, διότι το να ανταλλάσσουμε ποινικά μητρώα είναι, έχει νόημα για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια στους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι δικαίωμά τους. Ε, ε, από την εμπειρία μου ως Υπουργού Δικαιοσύνης ε, το 2004-2008 στην Ισπανική κυβέρνηση υιοθετήσαμε μια πρωτοβουλία όταν αυτή η υπόθεση ήταν ε, διακυβερνητική για να βάλουμε με αυτόματο και ηλεκτρονικό τρόπο μια διάταξη εξασφάλισης αυτής της δυνατότητας των κρατών μελών να ελέγξουν διασυνοριακά το ποινικά μητρώα και σε πλαίσια τα πολύ ευαίσθητα όπως είναι η εγκληματικότητα, η ε, σεξουαλική ε, εγκληματικότητα, ιδιαίτερα στα άτομα τα ιδιαίτερα ευάλωτα όπως είναι οι ε, ανήλικοι. Το κάναμε ανάμεσα στην Ιταλία, την Ισπανία, την Γερμανία, αν και μετά από λίγο η Ιταλία έφτιαξε ένα δικό της ε, σύστημα ε, και μετά βέβαια στη Λισαβόνα είδαμε ότι και είπαμε ότι θα έπρεπε αυτό να ε, ε, αναχθεί σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα με αυτή την μεγαλύτερη εγγύηση για ελευθερία όμως και ασφάλεια. Είναι λογική και σημαντική πρωτοβουλία και θα προσπαθήσω να συμβάλλω μέσω της κοιόδους της Σοσιαλιστικής Ομάδας στη σύνταξη τροπολογιών που θα τελειοποιήσουν την πρωτοβουλία της Κομισιόν και την πολύ λογική κατεύθυνση που υπέδειξε ότι θα ακολουθήσει ο συνάδελφός μας. Σας ευχαριστώ. Η, για την άλλη είναι η Σοφία Ιντφελτ, κοιόδης. Σας ευχαριστώ και εγώ θα είμαι σύντομη γιατί σε ένα λεπτό θα πρέπει να πάω σε μια άλλη συνεδρίαση όπου και προεδρεύω και είναι σε άλλο τμήμα του κτίριου. Συμφωνώ εκτενώς με την πρόταση του συζητητή και πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε κάποιες λεπτομέρειες ποιος θα καλύπτεται ακριβώς, τι θα γίνεται με τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διπλή υπηκότητα, και τους μη υπηκόους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι υπέρ της πρότασης μιας κεντρικής βάσης δεδομένων. Με βάση και ζωτάει όσα είδαμε προσφάτως με τη μη ανταλλαγή πληροφοριών, όχι μόνο σε περιπτώσεις τρομοκρατίας. Να κοιτάξουμε και τις προτάσεις σε ό,τι αφορά τη διαδικασία με την χρήση ψευδονύμων και όχι μόνο με την χρήση με Να δούμε και τις σχετικές αποφάσεις. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες και θα πρέπει να εξετάσουμε. Ε, συνολικά όμως ε, υποστηρίζω την γενικότερη κατεύθυνση την οποία προτείνει ο εισηγητής. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Γιάν Αλμπρέχτ από τους Πράσινους. Σας ευχαριστώ. Και εγώ γενικά υποστηρίζω την έκθεση και αυτά που προτείνει ο εισηγητής για την αντικατάσταση της ανωνυμοποίησης με τη χρήση ψευδονύμων. Σημαντική αλλαγή. Να τονίσω επίσης ότι καταρχάς θα πρέπει να ορίσουμε μία βάση hit, no hit. Αυτό φαίνεται ότι ισχύει. Επίσης, οι κατηγορίες δεδομένων που θα φυλάσσονται σε εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά καταδικασμένους Ευρωπαίους και μη Ευρωπαίους υπηκόους θα πρέπει να μην υπάρχουν διαφορές εκεί. Και τέλος, σε ό,τι αφορά τα δακτυλικά αποτυπώματα, θα πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει ένα εθελοντικό σύστημα για τα κράτη-μέλη, να μην καταστεί δηλαδή υποχρεωτικό. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή, λέει ο Πρόεδρος, εν συντομία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προφανώς και χαιρόμαστε ιδιαίτερα με την ευρεία υποστήριξη που λάβαμε από την Επιτροπή σας. Είναι καλή η πρόοδος της διαπραγματεύσης και προσβλέπουμε στη συνεργασία με το εισηγητή και τους κοιόδης και τώρα πάλι ο κύριος Κερκόπος, εισηγητής. Πρόεδρε, επικοδομητικός αυτός ο γύρος και νομίζω ότι σε τελική ανάλυση θα είναι πολύ καλή η συνεργασία για να πετύχουμε το σωστό κείμενο. Ελπίζω να μην μας πάρει τόσο πολύ αυτό το θέμα όπως ε, και σε άλλες περιπτώσεις εκθέσεων που έχω αναλάβει να μην μας πάρει 3-4-5 χρόνια και ελπίζουμε να μην ε, γίνει το ίδιο που έγινε στο PNR, να καταφέρουμε τέλο πάντων μέσα στη δική μου θητεία, τη δική σα θητεία, έστω, ε, Πρόεδρε, να το ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Τα λέμε το απόγευμα, λέει ο πρόεδρος.